Καλώς ήλθατε, καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε πρόβλημα με κάποιους συναδέλφους που δεν έχουν φτάσει ακόμη και δεδομένου ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Μαρία, ευχαριστώ που παίρνεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι εδώ στις 3 ε, και είναι σπάνιο. Βέβαια θα έκανα μια πρόταση για το μέλλον. Όταν έχουμε ψηφοφορίες, να μην τις βάζουμε 3 η ώρα τη Δευτέρα, γιατί ακόμη και την καλύτερη βουλή του κόσμου να έχουμε, κάποιοι δεν μπορούν. Εγώ ταξίδεψα χθε το βράδυ, γι' αυτό είμαι εδώ. Διαφορετικά δεν θα προλάβαινα αυτή τη ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν, να σημειώσει η γραμματεία για το μέλλον ότι να μην βάζουμε καθόλου ψηφοφορίες τη Δευτέρα, καλύτερα την Τρίτη. Ευχαριστώ. Πράγματι, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε συνήθω. Στην περίπτωση αυτή, όπω ξέρει, υπάρχει πρόβλημα με τι προθεσμίε, γιατί αύριο το απόγευμα θα ψηφίσει η Επιτροπή Περιβάλλοντο. Και μα το είχαν ζητήσει και άλλοι συνάδελφοι, επομένω αναγκαστήκαμε να θέσουμε τι ψηφοφορίε αυτέ ω πρώτο σημείο. Αλλά πιστεύω ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λεκού Κόμματο έφτασαν. Είχαμε κάποια προβλήματα με τα μέλη του ΕΛΚ. Νομίζω ότι τώρα είναι εδώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και ελπίζω να έρθουν και οι συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε όλοι λοιπόν. Εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από την πλευρά σας. Η ημερησία διάταξη για σήμερα και αύριο θεωρείται εγκεκριμένη. Να σας ενημερώσω ότι η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου και ότι έχουμε και διερμηνία σε 19 γλώσσες. Θα έλεγα λοιπόν να περάσουμε τώρα στο σημείο 3. Όπω γνωρίζετε, επιστηστική κρίση και η απάντηση στην τροφική και αντίστοιχη έλεγξη είναι το σημείο αυτό. Μιλάμε για ένα σχέδιο γνωμοδότηση τη κυρία Ουλρίκε Ρόντουστ. Όπως θα θυμάστε, στις 4 Νοεμβρίου είχαμε αρχίσει να εργαζόμαστε επί της έκθεσης Ρόντουστ, επί της έκθεσης Ιδίας Πρωτοβουλίας ε, για την επιστηστική κρίση, απάτη συντροφική αλυσίδα και αντίστοιχους ελέγχους. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι η αρμόδια επιτροπή. Η απόφαση για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετίζεται με το πρόσφατο σκάνδαλο που ανακαλύφθηκε σε ορισμένα κράτα-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει να κάνει με το κρέας αλόγου και αν θέλει και η κυρία Ρόντος να πάρει το λόγο θα μας το πει. Εδώ ζητούνται μέτρα για την αχνηλασιμότητα των τροφίμων και για να υπάρξει εγγύηση στο δικαίωμα ενημέρωση του καταναλωτή κατά της απάτης και ενίσχυσης των υγειονομικών κανόνων καθ' όλη την αλυσίδα παραγωγής. Έχουν κατατεθεί 73 τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Επομένως θέλω να ρωτήσω τον Ρίκη αν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που ε, εργάστηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τόσο εντατικά. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορούσαμε να έχουμε συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Αυτό συνέβη επειδή είχαμε τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Όμως σε όλες οι πολιτικές ομάδες, σε τεχνικό επίπεδο, συνεργάστηκαν στενά μεταξύ τους και επικοδομητικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ πολύ θερμά γι' αυτό και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Μακίνες ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοια ψηφοφορία τη Δευτέρα. Αλλά οφείλεται στο ότι βρισκόμαστε υποπίεση και αύριο η ΕΝΒΗ θέλει να ενημερωθεί σχετικά με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορέσαμε να, εργαστούμε, να συνεργαστούμε τόσο πολύ όσο στο παρελθόν, αλλά όλοι όσοι συνεργάστηκαν έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, έχουν προσπαθήσει πέρα από τα όρια των πολιτικών ομάδων να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ουλρίκε. Μπορούμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Έχετε όλοι την κάρτα σας. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ωραία, για να προσπαθήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τη συμβαστική τροπολογία 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Μένα ένα συγχυρός. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τώρα να περάσουμε στην τροπολογία 71 Σμιτ. Υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, είναι καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, ψηφίσατε όλοι. Δεν έχεις κάρτα. Λοιπόν, να λάβουμε υπόψη την ψήφο του κυρίου Λαβία. Ωραία. Εγκρίνεται θα έλεγα. Περνάμε στην τροπολογία 7. Άλβουρτ και λοιπή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία Νίκολσον. είναι 9. Ναι, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Νικολσόν υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Νικολέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη 14. Γκάμπριλ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Γιάρ. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 σκοτά, υπέρ, κατά, εποχέ, απορρίπτεται. 18 όσλινγκ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 Νίκολσον υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20. Σκοτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21. Χόσλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22. Σκοτά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 24 σκοτά υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται Τροπολογία 33. Γκαμπριέλ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια Ιούλη και Λιβύη 46, 38 μέχρι 46, με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 38-46. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Agreed. Περνάμε στις 47 με ένα χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα το μπλοκ 48 έως 50, Νίκολσον και Λυπή. υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 59 Νίκολσον υπέρ. Ψηφίζουμε την 59 υπέρ. Κατά. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. με ενημερώνουν ότι πρέπει να επιστρέψουμε και να ψηφίσουμε την 52 γιάρ. Ψηφίσουμε την 52 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά για την 52 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Θέλω ότι εγκρίνεται, αλλά ας δούμε. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 53 Νικουλέσκου. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται θα έλεγα. Είμαστε σίγουροι ή πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Ωραία, εγκρίνεται. 55. πέντε. Ρέιμερς υπέρ. Κατά. Εποχές υπορρίπτεται. Τώρα, 59, Νικουλέσκου. Νίκολσον, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος. 59, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται, θα έλεγα. Να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 59 Νίκολσον. Πέρας. Εγκρίνεται. 63 Reimers. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Μάλιστα. Για την 63 άρχεται η ψηφορία. Τροπολογία 63 Reimers. Ότι απορρίπτεται, ναι. Εγώ θεώρησα ότι με ευρία πλειοψηφία απορρίπτεται, αλλά μπορούμε να ελέγχουμε. Πέρας. Και όντως απορρίπτεται. Ξεκάθαρη ψήφος. Περνάμε τώρα στην 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Και εδώ νομίζω απορρίπτεται. τάση χειρό. 65 Νίκολσον υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 66 Μαγκίνες υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 67 Σμιθ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 67 Σμιτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Με εσύ χειρός. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται θα έλεγα. 73 ε, του εισηγητή. Της εισηγητρίας μάλλον υπέρ κατά προχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου έτσι όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια Ουλρίκη. Και μπορούμε τώρα να τα στείλουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να λάβουν υπόψη και τη δική μας νομοδότηση. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερησία διάταξης. Πρόκειται και εδώ για μια γνωμοδότηση που κατόπιν ε, της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων ε, των κρατών μελών στην Κομισιόν είναι πολύ σημαντική. Όπως ε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μπορείτε να δείτε στην Ολομέλεια οι εκτελεστικές και κατεξοδότητες πράξεις που σχετίζονται με τη γεωργική νομοθεσία μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για το ζήτημα αυτό λοιπόν ψηφίζουμε σήμερα μία έκθεση πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων που είναι η αρμόδια επιτροπή όπως ξέρετε έχει εδώ κατατεθεί μόνο μία τροπολογία της κυρίας Λούλινγκ ε, που ζητά από την Επιτροπή να μην καταχραστεί της κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα έλεγα να ψηφίσουμε τη μοναδική τροπολογία της κυρίας Λούλινγκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πρέπει να έχουμε και μια τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία για το τελικό κείμενο της γνωμοδότησης, ηλεκτρονικά. Πέρας. Και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, 24 προς 3. Ευχαριστώ. Υπάρχει ακόμα μία ψηφοφορία. Σημείο 5 της ημερησής διάταξης. Πρόκειται για ένα μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ ε, της Αμερικής το έχουμε ήδη συζητήσει και αφορά την εισαγωγή βοηού κρέατο από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένε αυξητικέ ορμόνε και σχετικά με του αυξημένου δεσμού που επιβάλλονται από τη ΣΥΠΑ σε ορισμένα προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ βιαζόμαστε γιατί η αρμόδια επιτροπή είναι η επιτροπή ΙΝΤΑ Διεθνού Εμπορίου που θα πρέπει να ψηφίσει στι 27 του μήνα. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση και είμαι εγώ ο εισηγητής σε σχέση με το αναθερμένο μνημόνιο συμφωνία με τι ΗΠΑ για την εισαγωγή βιοκρέατο υψηλή ποιότητα. Και καθώς πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν τροπολογίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε εδώ τη διαδικασία της συνένεσης. Μπορούμε απλώς ε, να δεκτούμε ή να απορρίψουμε το κείμενο. Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο κύριε Μποβέ. Πρόεδρε, μια ερώτηση. Δεν κατανοώ γιατί στα προσψήφιση έχουμε προβλέψει ένα θεώρηση κάθε 6 μήνες. Γιατί όχι κάθε ένα χρόνο. Δεν βλέπω την αναγκαιότητα αυτής της δυνατότητας συνεθεώρησης κάθε έξι μήνες. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, Είναι διαδικαστικό το θέμα, Ζωζέ, όπως μου εξηγεί τώρα η γραμματεία. Γιατί αν δεν προβαίναμε σε ψηφοφορία, απλώς θα κατέπτυπτε αυτή η διαδικασία η εξεμηνέα. Έτσι λοιπόν με την ψηφοφορία αυτή επιτρέπουμε τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Είναι λοιπόν αναγκαιότητα αυτό προκειμένου να υπάρξει αυτός ο έλεγχος. Πρέπει μόνο να ψηφίσουμε λοιπόν αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Ναι ή όχι. Λουίς. Τζοζέ και πάλι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Το ότι πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ναι, το να περάσουμε από τη φάση 2 στην 3, σύμφωνοι. Και το υποστηρίζω. Διότι βγαίνουμε από μια μάχη, η οποία κράτησε 12 χρόνια και είμαστε πλέον στην τελική διαπραγμάτευση. Μέχρι εδώ καλά. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί το εξάμεινο αυτό, τη σχετική πρόβλεψη, την προσθέτουμε εδώ. Που θα επιτρέψει δηλαδή στις ΗΠΑ να αναπροσαρμόζουν τις εισαγωγές με τέτοια συχνότητα. Να κλείνουν την στρόφη κατά τη στιγμή που προχωρούμε προς μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Γιατί κάνουμε αυτό το δώρο λοιπόν στους ε, οικονομικούς μας εταίρους μου επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια διαδικασία ζωζέ εντελώ συνηθισμένη, γιατί αν δεν ψηφίσουμε τότε δεν θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να έχει αυτό το δικαίωμα για τον εξεμηνίο έλεγχο. Είναι μια συνήθις πρακτική. Αν κατόπιν θέλεις να το δούμε το θέμα εις βάθος, ίσως ε, εν ευθέτω χρόνο. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Πρέπει να έχουμε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία υπέρ, κατά. Votazione Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Περνάμε τώρα σε ένα θέμα προβληματισμού Σημείο 6. Υγεία των ζώων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Πόλσεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Τώρα θα ξεκινήσουμε και την ακρόαση για την ευημερία των ζώων και θα μπορέσουμε να ακούσουμε και τους εμπειρογνώμονες και τα ενδιαφερόμενα μέρη για το θέμα αυτό. Αλλά καταρχήν θα ήθελα να καλέσω την εισηγήτρια να παρουσιάσει την εκθεσή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για έναν κανονισμό σχετικά με την υγεία των ζώων αποσκοπεί στην αντικατάσταση 40 περίπου διαφορετικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα αυτών, εκ των οποίων η παλαιότερη χρονολογείται από το 1964. στόχος είναι να θεσπίσουμε ένα ενιαίο πλουστευμένο, διαφανές και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο που θα καθιστά δυνατή μια ξεκάθαρη και ισορροπημένη κατανομή καθηκόντων και ευθυνών σε σχέση με την παρακολούθηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των διαφόρων ε, μεταδοτικών νόσων των ζώων. Η πρόταση της ε, Επιτροπής έχει τεράστια σημασία και για τη δημόσια υγεία, καθότι το 70% των μολυσματικών ασθενειών που μας πλήττουν είναι κοινέ στα ζώα και στους ανθρώπους. Η πρόταση όμως ε, δεν αφορά μια νομοθετική πράξη για την υγεία των ζώων καθ' αυτή. Περισσότερο έχει να κάνει με τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων. Στόχος είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή από τα ζώα στον άνθρωπο. Ένας Ευρωπαϊκός Νόμος Προστασίας των Ζώων, ο οποίος θα περιέχει γενικές αρχές σχετικά με το καθήκον της μέρημνας και την κατανομή ευθυνών και εκπαιδευτικών απαιτήσεων, θα ήταν ιδιαίτερος χρήσιμος για τους αγρότες και τα ζώα στην Ευρώπη. Και είναι κάτι που έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, αυτό που προτείνει σήμερα η Επιτροπή διαφέρει εντελώς από κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η καλή μεταχείριση των ζώων είναι άσχετη με το θέμα. Αντιθέτως, υπάρχει αδιαμφισβήτητη αλληλουχία μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των ζώων και των ανθρώπων. Αυτή είναι μια κέρια επιλογή προσέγγισης, η οποία ονομάζεται One Health, μία υγεία και η οποία ευτυχώς αντανακλάται στο άρθρο 10 της πρότασης. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πράξη να διέπεται από αυτή την προσέγγιση και να εξερνίζεται τη σύνδεση μεταξύ ορθών ζωοτεχνικών πρακτικών και καλής υγείας των ζώων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι τα αδέσποτα ζώα και αυτά μπορούν να γίνουν αιτία διάδοση σε λιμωδών νόσων. Απαιτούνται ισχυρά μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Τα δέσποτα είναι λίγο πολύ το ίδιο με τα άγρια ζώα. Ε, δηλαδή ε, ζώα τα οποία δεν έχουν έναν υπεύθυνο ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με την πρόταση, θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσία να συμπληρώνει το περιεχόμενο του κανονισμού με 106 κατεξουδότηση πράξη και 57 εκτελεστικέ ε, πράξει. Σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα, η οποία προβλέπει περίπου 600 περιπτώσεις των λεγόμενων διαδικασιών επιτροπολογίας, πρόκειται προφανώς για θετική εξέλιξη. Όμως ε, πρέπει να αλεχθεί ότι μόνο οι μισές περίπου από τις προτινόμενες και εκτελεστικές πράξεις πράγματι αυξάνουν τις σημερινές εξουσίες της Επιτροπής. Ε, τα περισσότερα δηλαδή στοιχεία εδώ ήδη υπάρχουν. Σημαντικό είναι να μπορεί να τροποποιηθεί γρήγορα ο κανονισμός, ε, για παράδειγμα σε περίπτωση ε, επιδημίας. ή σε περίπτωση εμφάνισης μιας νέας νόσου. Και δεν έχει νόημα να νομοθετούν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της παραμικρής λεπτομέρειας ε, στον, ε, στο πολύπλοκο αυτό σύστημα ε, κανόνων. Χρειάζεται να βρεθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ προβλέψιμότητας και ευελιξίας. Είναι σημαντικό το κείμενο του κανονισμού να περιέχει τις βασικές αρχές και κατευθυντήρες γραμμές. Οι λεπτομέρειες ε, μπορούν κάλλιστα να συμπληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους επιρογνώμονές τη ε, σε ε, μεταγενέστερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση, οι αποφάσεις της Επιτροπής να με βάση τα πιο αξιόπιστα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και γνώσεις. Επίσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική αναφορά 13 της πρότασης της Επιτροπής, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων. Γενικά πάντως μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, αυτή είναι σαν να αγοράζουμε γουρούνι στο σακί. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν στην πράξη αύριο όλες αυτές οι διατάξεις και ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεωθεί τουλάχιστον στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αυτή η έκθεση θα πρέπει να περιέχει ανασκόπηση της αποκομιστής ασπίρας από την εφαρμογή του κανονισμού και των πρόσθετων νομικών πράξεων που εγκρίθηκαν. Και εφόσον είναι σκόπιμο, να συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις. Άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της πρότασης αυτής είναι η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνεται στην ταχεία λήψη αποτελεσματικών μέτρων με στόχο τον έλεγχο και την εκρίζωση ορισμών ασθενειών. Κάτι που είναι και χρήσιμο και ευπρόσδεκτο. Όμως, το μεγαλύτερο κόστος για την κοινωνία και για τους γεωργούς μας ε, ε, το επιφέρουν οι ε, εντυμικές ασθένειες που δεν θα αναφέρονται στον κανονισμό αυτό. Τέτοιου τύπου ασθένειες αντιμετωπίζονται εν μέρη με αντιβιωτικά. Σχετίζονται συνεπώς με το διαρκώς διευρυνόμενο πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο κανονισμός αυτός να περιέχει και απαιτήσει σε περί προληπτικών προορατικών μέτρων παρακολούθησης και ελέγχου και αυτών των μη καταγραφόμενων ασθενειών, ακόμα και αν αυτό θα πραγματοποιείται σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης έχουμε ένα άλλο πρόβλημα σημαντικό. Θέλουμε ελεύθερη αγορά, αλλά όχι ελεύθερη διάδοση των ασθενειών. Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κέρια σημασία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κανείς φαντάζομαι δεν νοσταλγεί τις ημέρες των συνοριακών ελέγχων. Κάποια κράτη-μέλη και περιφέρειες όμως έχουν ε, καταφέρει με πιο αποτελεσματικό τρόπο να εκριζώσουν ασθένειες ε, στο έδαφος τους. Ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει λοιπόν ε, κάποιο τύπο ισορροπία. Θα πρέπει να επιτρέπονται μέτρα προστασίας, αλλά υπό την προϋπόθεση να βασίζονται σε αυστηρά επιστημονική βάση και να μην εγκρίνονται για οικονομικούς λόγους για να λειτουργήσουν ως συγκεκαλυμμένοι περιορισμοί στο εμπόριο. Θέλουμε ελεύθερη αγορά, όχι όμως ελεύθερη διάδοση ε, των ασθενειών. Σας ευχαριστώ. Molto bene, grazie. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο Πόλσεν για την παρουσίαση αυτή. Τώρα, το πρόγραμμα είναι το εξή. Θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου που το επιθυμούν. Κατόπιν θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη ΓΑΜΑ ΔΑΛΤΑ ΣΑΝΚΟ, τον διευθυντή Βαν Γκίτεν, που είναι παρόν. Και στη συνέχεια θα περάσουμε και στην ακρόαση. Θα ζητήσω και από του εμπειρογνώμονε να έρθουν εδώ στο βήμα τον καθηγητή Βάξο και την ε, κυρία συγγνώμη και τον κύριο Βαλεντίνο Αλμάσα Δελάρα ο κύριος Άγνιου καταρχήν παρακαλώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Με εκπλήσει κάπως που μου δίνετε εμένα πρώτο τον λόγο. Κάποιες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω ε, σε απάντηση στην ε, κυρία ε, Πόλσον. Λέει ότι κανείς δεν νοσταλγεί τις ένδοξες μέρες των συνοριακών ελέγχων. Εγώ τις νοσταλγώ και σκέφτομαι ιδιαίτερα τη Λίσα. Λίσα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχαμε πει πολλά χρόνια. Εξαπλώνεται τώρα όμως προς τις ακτές μας από την Ανατολική Ευρώπη μεταδίδεται ε, συνεχώς και είναι σοβαρή ασθένεια και για τα ε, σκυλιά και για ε, το, τους ανθρώπους. Ε, εγώ θα ήθελα λοιπόν να είμαι απολύτως βέβαιος ότι κανείς δεν κρύβει στις αποσκευές του σκύλο άρρωστο. Και το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ο αφρικανικός πυρετός των χείρων. και είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται προς τα δυτικά από την Ασία. Στη χώρα μας έχουμε αναπτύξει ε, θεραπεία για την ασθένεια. Αυτό μπράβο λοιπόν στους Βρετανούς επιστήμονες, ωστόσο έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ε, ε, ε, ε γενετική τροποποίηση για να το κάνουν αυτό και δεν τους επιτρέπεται να προχωρήσουν αυτή τη θεραπεία λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του πράσινου του οικολογικού λόμπι. και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε σήμερα να ακούσουμε μια απάντηση σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άγνιου. Ελίζαβετ Γέγγελ και κατόπιν ε, Σμιτ. Παρακαλώ Ελίζαβετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσον για τη δουλειά που έχει κάνει ε, σε σχετικά, χρονικό, σε, σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για ένα πολύ ευρύ θέμα. Διότι ε, ε, ε, όποιος γνωρίζει πόσα καλύπτει η έκθεση αυτή, πόσα, πρέπει να, πόσα πράγματα πρέπει να προσέξει, να διαβάσει, να μελετήσει, ε, θα διαπιστώσει ότι και σε καλή συνεργασία με άλλους ε, έχει υποβάλει μια πολύ καλή πρόταση. Ε, θα ήθελα να τονίσω όλα τα επιμέρους σημεία που ανέφερε. Περιμένω εναγωνίως να δω τι μπορούμε να μάθουμε από την σημερινή ακρόαση. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι μία πρόταση για την υγεία των ζώων και όχι για την ε, καλή διαβίωση των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε να κάνουμε τη διάκριση αυτή. Τα σημεία που ανέφερε η κυρία Πόλσεν, αυτά να τονίσουμε και όχι άλλα, τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα. Καταλαβαίνω τον κύριο Άγνιου. Από την άλλη όμως ζούμε τώρα πια σε έναν κόσμο ανοιχτό που έχει ανοιχτά σύνορα. Και μιλάμε μεν για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν χρειάζεται καν να κρύψει κάποιο πρόσωπο ένα σκύλο στις αποσκευές του και ο αέρας μεταφέρει ασθένειες τώρα πια. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε μια λογική αντιμετώπιση που να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα λύσας, ε, ε, ε, υπάρχει και με υπάρχει και με, τους ασβούς, γι' αυτό δεν έχει νόημα μια τέτοια αντιμετώπιση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την ε, κυρία Πόλσεν, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους ε, που έχουν συνεργαστεί στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ελίζαμπετ. Παρακαλώ, συνάδελφος Μίτ. Θα είμαι πολύ σύντομο ως συζητητής ε, για την ομάδα μου και θα ήθελα να συμπληρώσω την τα σχόλια. Συγχαίρω την κυρία Πόλσεν ε, για την προσέγγιση που ακολουθεί στην έκθεση αυτή και συμφωνούμε που εστιάζεται στις ε, μολυσματικές ασθένειες. Ε, νομίζω ότι υπάρχει και ένας πειρασμός και για άλλους βουλευτές από άλλες επιτροπές να θέσουν και άλλα ζητήματα εντός της έκθεσης. Όμως εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ να είμαστε κάπως πειθαρχημένοι για να δούμε πού θέλουμε να φτάσουμε. Επίσης, συγχαίρω την κυρία Πόλσεν για τόσο αναφέρει για την ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και κατοξιότητας πράξεων και θα ήθελα να ακούσω και την Κομισιόν πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στο θέμα αυτό. Όμως, σήμερα θέλουμε να ακούσουμε και άλλους ομιλητές, έτσι λοιπόν εγώ δεν θα μακρηγορήσω. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Τώρα, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ, στον Διευθυντή Μπέρναρτ Βαν Γκίτεν. Παρακαλώ. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ την κυρία Πόλσον για την τεράστια δουλειά που έκανε. Το είπε και η ίδια. Τεράστια δουλειά καταργούνται τέσσερις οδηγίες που διέπουν τον τομέα και στο οποίο βαριστήκαμε τα τελευταία 50 χρόνια. Τις 600 νομοθετικές πράξεις που χρειαζόμασταν κατόρθωσαν τις περιορίσει σε 260. Και απλούστευση, λοιπόν. Όμως απλούστευση δεν σημαίνει ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με εξάπλωση των ασθενειών. Αυτός μην το ξεχνούμε. Ακούσαμε για την λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξαπλωσή της. Θυμίζω όμως τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο τα κρατη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισαν τις ασθένειες και τις περιόρισαν σε συγκεκριμένες περιοχές τα τελευταία χρόνια. Θυμηθείτε τον αυθόδη πυρετό το 2001. Τα καταφέραμε χάρη ακριβώς στην περιφερειοποίηση, στην λήψη περιοριστικών μέτρων. Αυτή είναι την προσέγγιση ούτως ή άλλως υιοθετούμε εδώ και πολλά χρόνια. Η τακτική μας είναι λοιπόν να περιορίζουμε τις ασθένειες εκεί που εκδηλώνονται. Το σύνθημα νομοδότησης συνάδει με τις προτάσεις μας επί της ουσίας όσον αφορά την κεντρική ιδέα αν θέλετε και εννοείται ότι δεν αφορά ούτε τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ούτε την προστασία των ζώων. Αφορά τις ζωονόσους. Και τα μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε αναπαραγωγή χωρίς ασθένειες. Για να μην έχουμε θέματα δημόσιας ε, υγείας ή ασφαλείας. Οι κανόνες στην υγεία των ζώων είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, όταν τα κρατημέλη καλούνται να αντιμετωπίσουν ε, συγκεκριμένες ασθένειες, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει και η κοινωτική διάσταση. Γι' αυτό και δεν θέλουμε τα κράτη-μέλη με δική τους πρωτοβουλία να διατεράσουν την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όσον αφορά τη κατεξουδότηση και τις εφαρμοστικές πράξεις, όπως ήδη είπαν διάφοροι προλαλήσαντες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να έχει την δυνατότητα να θεσπίζει νομοθεσία επί σειράς θεμάτων σε στενή συνεργασία βεβαίω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κρατη Το τελευταίο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι αυτό το οποίο έφτιαξε η κυρία Πόλσεν στην αρχή της ομιλίας της. Τα αδέσποτα σκυλιά που είναι πρόβλημα σε ορισμένες χώρες καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία η οποία επιτρέπει ακριβώς να λαμβάνονται μέτρα βάσει της φυστάμενης νομικής ε, βάσης για τον περιορισμό των δεσποτών σκύλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Γενική Διεύθυνση Σάνκο και θα ξαναδώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο Πόλσεν πριν να δώσουμε το λόγο στην περιεχόμενη. Παρακαλώ, Μάρη. Ναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά την ε, Βρετανική θέση. Κι εγώ Σουηδέζα είμαι. Και υπάρχει σημαντική πίεση στην πατρίδα μου να διατηρήσουμε τη, τους ελέγχους στα σύνορα, στα σύνορα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία σε σχέση με την ανάγκη μας να έχουμε μια αγορά που να λειτουργεί καλά. Ε, βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης με πολύ ψηλή ανεργία. Ε, χρειαζόμαστε ε, μια δυναμική οικονομία. Αλλά στην πρότασή μου υπάρχουν και ειδικές προϋποθέσεις για τα κράτη-μέλη που έχουν σύνορα με την Ανατολική Ευρώπη. Να ε, λάβουν, για παράδειγμα, ειδική επιχορήγηση για την καταπολέμηση ε, της πανόλης των χείρων. Είναι σημαντικό αυτό, νομίζω όμως ότι πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Όσον αφορά τις κατεξοδιώτες πράξεις, στην παρούσα πρόταση υπάρχει κάπως πιο αυστηρή διατύπωση σχετικά με το πώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν ε, της, τη, γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων και των επιστημόνων κατά την εκπόνηση των κατευθυντών πράξεων. Επίσης, η Κομισιόν σε πέντε χρόνια από τώρα θα πρέπει να υποβάλει ανασκόπηση των όσων έχει καταφέρει και το πώς λειτουργούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πόλσεν. Η κυρία Πέρες έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη ερώτηση θέλω να κάνω, καθώς άκουσα τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Κάποια συγκεκριμένη στιγμή αναφέρθηκε σε κάποια άγρια ζώα. Είναι ένα θέμα που ήθελα να το θέσω μέσω της κατάθεσης τροπολογιών, αλλά ήδη υποφελούμε της ευκαιρίας που μου δίνεται εδώ. Υπάρχει στην οδηγία αυτή η έννοια των άγριων ζώων και δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα ερμηνείας μόνο στα ισπανικά, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε ένα διαφορετικό όρο αντί για σαλβάχε να λέμε Σιλβέστρες στα Ισπανικά, γιατί ε, έχουμε παραδείγματο χάρη πολλές φορές τις αγελάδες που βόσκουν ελεύθερα, δεν είναι άγρια ζώα όμως έτσι λοιπόν τώρα κάθε φορά που στο κείμενο αναφέρεται ο όρος ε, σαλβάχε θα έπρεπε να αλλάξει και να λέμε σιλβέστρια άγρια ζώα. Bene, eh, να απαντήσει. Μπορώ να σου απαντήσω. Ο ορισμός των αγρίων ζώων είναι τα ζώα που δεν έχουν ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή κάποια εταιρεία που να έχει την ευθύνη για το ζώο αυτό. Νομίζω ότι είναι ο σαφέστερος ορισμός που μπορούμε να έχουμε. Εάν δηλαδή έχουμε ένα σκύλο χωρίς ιδιοκτήτη που ζει στο δρόμο ή ε, ε, εάν έχουμε ένα ζώο στο δάσος το θέμα είναι το ίδιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά επιμένω ότι πρόκειται για ένα θέμα γλωσσικό και ερμηνεία τουλάχιστον στα ισπανικά, στα καστιλιάνικα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με είπε η κυρία Πόλσεν, όμω το κείμενο στα ισπανικά λέει animal salvaje και ένα εγκαταλειμμένο σκύλο δεν είναι άγριο ζώο. Επομένως, εγώ συμφωνώ μας λέει η κυρία Πόλσεν, ε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα και σε άλλες γλωσσικές εκδοχές. Πρόεδρος, Κομισιόν παρακαλώ, θέλετε το λόγο. I'm sorry, Mr. Chairman, my... Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Τα ισπανικά μου είναι ελαχιστότητα. Κυρία Πόλσεν, κατανόησε, είμαι βέβαια στο πρόβλημα. Εμείς αναφερόμαστε τα ζώα τα οποία ζουν ελεύθερα στη φύση. Απλώς. Μάλιστα, θα διερευνήσουμε το ζήτημα. Ευχαριστώ. Και συνεχίζω ο πρόεδρος στο μικρόφωνο. Μάλιστα, θα έλεγα μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ακρόση, δίνοντας καταρχήν το λόγο στους δύο προγνώμονες που βρίσκονται εδώ στο βήμα της Προεδρίας, τον κύριο Ιβαρ Βάξον, καθηγητή στο Συνδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονίας και κατόπιν στον κύριο Βαλεντίν Αλμάν Σαδελάρα, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας της Ισπανίας. Έχετε από 10 λεπτά ο καθένας. Και κατόπιν θα περάσουμε στη συζήτηση, αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ με τέσσερις ακόμη ομιλητές. Παρακαλώ, οι εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ σήμερα και ε, ζητώ συγγνώμη που <laughs> έχω λίγο τρακ. Νομίζω ότι θα ήθελα να ξεκινήσω από την πρόταση αυτή. Ως επιστήμον, έχω ε, συμμετάσχει σε επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και 16 χρόνια. Εγώ ως μη νομικός κρίνω ότι η δουλειά αυτή είναι αρκετά καλή που έχει γίνει. Αλλά εδώ έχουμε έναν ε, νόμο για τις μεταδοτικές ασθένειες των ζώων, ε, όχι για την υγεία των ζώων. Καλύπτει κάποιες μεταδοτικές ασθένειες ε, όπως είναι ο φθόδης η κλασική πανάλη των χείρων. Ενώ ε, απλές ασθένειες όπως είναι η διάρκεια για παράδειγμα στα ζώα δεν καλύπτεται. Κάτι Άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι κάποια στιγμή θα χρειαστούμε ένα νόμο για την υγεία των ζώων και μάλλον σχετικά σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι καλή ε, επιστημονική βάση για κάτι τέτοιο μάλλον δημιουργείται αυτή τη στιγμή με τη χρήση ε, δικτών ε, καλής διαβίωσης των ζώων. Και η τρίτη μου παρατήρηση που νομίζω θα τη στηρίξουν και άλλοι ομιλητές είναι ότι η ε, ελεύθερη κινητικότητα για τα ζώα δεν θα πρέπει να σημαίνει και ελεύθερη μετάδοση των ασθενειών. Και νομίζω ότι ακριβώς κάτι τέτοιο προσπαθεί να πετύχει ε, η παρούσα νομοθετική πράξη. Εάν δεν ελέγξουμε τις ε, ασθένειες των ζώων, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μία ε, αγορά για ζώα και ε, ζωικά προϊόντα που να λειτουργεί καλά. Αποτελεί δηλαδή προϋπόθεση για την εσωτερική αγορά κάτι τέτοιο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, προσπάθησα να κοιτάξω τις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες ε, Μιλάμε λοιπόν για το γουρούνι στο σακί. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι μορφή τελικά θα έχει ε, αυτή ε, η νομοθετική πράξη και είτε μιλάμε για γουρούνι στο σακί είτε μιλάμε για γατί στο σακί ανάλογα με τη γλώσσα. Ε, φαντάζομαι ότι οι μεταφραστές μπορούν να με βοηθήσουν ε, αλλά ε, είναι πολύ χρήσιμο το να έχουμε επανεξέταση της νομοθεσίας αυτής μετά από πέντε χρόνια εφαρμογής. Κάτι που ανέφερε η εισηγήτρια είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα δεδομένα σε επιστημονικά δεδομένα. Και νομίζω ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς να έχει επιστημονικά στοιχεία στα οποία να βασίζει τις ε, προτάσεις ε, νομοθεσίας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ε, μπορούμε να δημιουργούμε νομοθεσία ε, που να μπορεί να εφαρμοστεί για πολλά χρόνια. Επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι η καλή διαβίωση των ζώων και η καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των ζώων ε, συνδέονται στενά μεταξύ τους. Εάν θέλουμε καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να έχουμε και υγεία, καλή υγεία των ζώων. Ε, χάρηκα πάρα πολύ που ε, σε σχέση με τις ε, στρατηγικές εκρίζωσης των ασθενειών αναφέρθηκε και η καλή διαβίωση των ζώων. Εγώ χαίρομαι όταν διαβάζω αυτή την νομοθετική πρόταση. Επίσης θα ήθελα να πω ότι όπως θα σημειώσετε και αρκετοί άλλοι ομιλητές, όσον αφορά το θέμα της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά, είναι κάτι που μας ε, χαλάει τη, τη γιορτή κατά κάποιο τρόπο. Ε, ε, και δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι η προορατική προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα ζώα ε, εκτροφής, αυτά που μπορούν να μεταδώσουν ε, την, ε, τα ζώα αναπαραγωγής. νομίζω ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο να επικεντρωθούμε σε αυτά παρά στα σφάγια. Θα ήθελα να Αναγνωρίζω τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών ε, σήμερα. Υπάρχουν ε, αρκετές ιστορίες επιτυχίας την τελευταία 20 ετία. Και θα ήθελα να πω ότι η ε, εκρίζωση της ΣΕΒ ή της Σαλμονέλας είναι περιπτώσεις που δείχνουν τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κάπως πιο εύθραυστη και μάλιστα αντιστρέψει μπορεί να είναι ε, η ε, ε, προσπάθεια ελέγχου της σαλμονέλας στα αυγά και στα πουλερικά. Θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε μια παρόμοια ιστορία επιτυχίας στον τομέα της ανθεκτικότητας των αντιβιωτικών, διότι σε κάποια κράτη-μέλη τώρα βλέπουμε ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, στο μισό των σφαγίων των, των κοτόπουλων. Ε, και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Υπόθηκε και νομίζω ότι θα επαναληφθεί αρκετές φορές ε, σήμερα. Ε, τα ε, υγιή ζώα δεν χρειάζονται αντιβιωτικά. Θα πρέπει σε ένα νόμο περί υγείας των ζώων να εισάγουμε τα στοιχεία αυτά που μπορούν ε, να βοηθήσουν στον έλεγχο της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά και ελέγχοντας ε, τα ζώα ε, που πολλούνται και τα ζώα αναπαραγωγής θα πρέπει να κοιτάξουμε την βιοσφάλεια στα, στις ενεργοτικές εκμεταλλεύσεις και γενικά τις καλές πρακτικές. Είναι δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός των αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται, ε, που φαίνεται από την απαγόρευση τη Ευρωπαϊκής Ένωση για την ζωοτεχνική χρήση αντιβιωτικών ε, στη ζωική παραγωγή. Ε, επίσης έχουμε ένα παράδειγμα από την Ορβηγία πριν από πολλά χρόνια στην παραγωγή σολομού. Όταν ξεκίνησα την σταδιοδρομία μου πριν πολλά χρόνια, η παραγωγή ανερχόταν σε 80.000 τόνους το χρόνο και η κατανάλωση αντιβιωτικών ε, ε, ανερχόταν σε 40 τόνους. Ε, το, σήμερα, 25 χρόνια μετά, η κατανάλωση αντιβιωτικών ανέρχεται σε 40 κιλά, δηλαδή μείωση κατά 9 ε, τα 100, ενώ η παραγωγή σολομού ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο τόνους, ε, δηλαδή 10 ε, φορές υψηλότερη. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι κατά την εκπόνηση μιας τέτοιας νομοθετικής πράξης νομίζω μπορεί να νιώθει κανείς περήφανος όσο όταν έχει συνορμολογήσει ένα επιπλοϊκέα είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα πετύχουμε. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για ε, ελεύθερη μετακίνηση των ζώων ε, δεν θα πρέπει να μιλάμε για ελεύθερη διάδοση των ασθενειών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στα ζώα αναπαραγωγής και χρειαζόμαστε ε, μια ιστορία επιτυχίας παρόμοια με άλλες που είχαμε στο παρελθόν ε, στον τομέα της, ανθεκτικότητας, ε, της καταπολέμησης ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βόξχολμ. βρίσκεστε καθοδόν προς την Εύσα, στην Πάρμα, όπου θα εργαστεί τόσο εμπειρογνώμονας. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο Βαλεντίν Αλμάνσα. από το Υπουργείο Γεωργίας ε, της Ισπανίας. Παρακαλώ. Ε, <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση στην ακρόαση αυτή και για την δυνατότητα που μας δίνεται να εκθέσουμε μια πολύ γενική άποψη του Υπουργείου Γεωργίας εν ώψη μιας τέτοιας πολύπλοκης ε, πρότασης. Ε, βρισκόμαστε σε νέους καιρούς, ε, ήδη είχε καθοριστεί σε ένα έγγραφο που συζητήσαμε πριν καιρό ότι καλύτερα η πρόληψη παρά η θεραπεία. Βρισκόμαστε σε ένα κόσμο που όλα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα στα πλαίσια της μεκοσμοποίησης και έχουμε και νέες αναδυόμενες νόσους. Ε, μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για και για άλλα ζητήματα και επομένω, χρειάζονται νέα εργαλεία. Και γι' αυτό η Κομισιόν αυτό που μα θέτει ε, είναι ένα νέο εργαλείο που πιστεύουμε ότι είναι καλά συντονισμένο στο τμήμα ενό ε, ευρύτερου πακέτου, πιο συνολικό, ότι ευθυγραμμίζεται καλύτερα με του ε, διεθνεί κανόνε, με το Διεθνές Γραφείο Πιζοποιών. Πιστεύουμε ότι είναι πιο απλή η νομοθεσία αυτή και πιο ευέλικτη. Επομένω, πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά θετικά σε αυτή τη νέα πρόταση τη Κομισιόν. Αυτό που μας αρέσει περισσότερο είναι να διατηρήσουμε στο επίκεντρο την υγεία των ζώων. Για μας είναι θεμελιώδες όμως ε, θα μου επιτρέψετε να ε, αναφερθώ και σε πράγματα που δεν μας αρέσουν και τόσο πολύ. Ένα από τα προβλήματα της ε, πρότασης είναι και μία από τις επιτυχίες της, ότι είναι υπερβολικά γενική η Κομισιόν αυτό που υιοθέτησε είναι η απόφαση να αποκτήσει πολλές αρμοδιότητες, πολλές εξουσίες. Καλό αυτό μένει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν ε, μπορούμε σε όλα τα άρθρα να συναντάμε δύο ή τρεις ε, φορές ε, της κατεξουσιοδότηση πράξης πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν η πρόταση και θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να μείνουν στην βασική νομοθεσία και κάποια θέματα που πρέπει να είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να είναι αρμόδια η Κομισιόν, αλλά ίσως για κάπως λιγότερο επίσης. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο σε ορισμένες περιπτώσεις να αξιολογήσουμε την πρόταση, γιατί είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τους κανόνες ε, για ορισμένες ασθένειες, όταν δεν ξέρουμε για ποιες ασθένειες, για ποιες νόσους μιλάμε, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλογοι. Έτσι λοιπόν, ε, πώς ε, θα πούμε αν το μέτρο Χ είναι κατάλληλο για μία νόσο που δεν γνωρίζω, πρέπει να ξέρω πρώτα τι νόσο. Έτσι λοιπόν, αυτή η γενικότητα ή μας καθιστά δύσκολο να ξέρουμε πού οδεύει η πρόταση σε ορισμένες περιπτώσεις. Ε, και για να συνεχίσω με τα επιχειρηματά μου, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αφήσουμε στο βασικό κανονισμό Ορισμένα σημαντικά θέματα, εδώ συμφωνούμε με την εισηγήτρια του Κοινοβουλίου, Δηλαδή τουλάχιστον ο νόσος, ε, το, μάλλον ο κατάλογος των νόσων προτεραιότητας ε, και η κατηγοριοποίηση των νόσων θα πρέπει να μείνει στο βασικό κανονισμό, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα θέματα αυτά εκ των προτέρων για να μπορούμε να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και ποια ζώα πλήττουν, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και κάποια συστήματα που θα μας επιτρέπουν πολύ γρήγορα να πούμε τους καταλόγους. Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά ο πρώτος κατάλογος πρέπει να μείνει στον κανονισμό. Επίση πιστεύουμε ότι το άρθρο 8, που είναι ένα καλό άρθρο, μπορεί να πλουστευτεί περισσότερο και να αποσαφινιστεί, γιατί όπως είναι η διατύπωση σήμερα, δεν ε, μας δίνει μια σαφή σύνδεση μεταξύ της νόσου και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για κάθε νόσο. Είναι λοιπόν δύσκολο να ερμηνευτεί το άρθρο αυτό και πιστεύουμε ότι η τροπολογία της κυρίας Πόλσεν βελτιώνει το κείμενο, αν και θεωρούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και να είναι πιο σαφές το κείμενο. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι απαραίτητο να μην ξεφύγει η κατάσταση από τα χέρια μας. Υπάρχουν κάποιες ε, νόσοι που δεν χρειάζονται τόσα μέτρα ελέγχου. Πρέπει να μην υπερβάλλουμε, δηλαδή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούμε να προσαρμόσουμε την αντίδρασή μας ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι πραγματικά η νόσος. Και το δεύτερο μεγάλο στοιχείο, κύριο στοιχείο, είναι το εξή. Κάποια πράγματα πρέπει να είναι στο βασικό κανονισμό και κάποια άλλα πράγματα θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ε, αποφάσεις ε, και να μπορούν να αξιολογούν τα μέτρα που είναι πιο κατάλληλα ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε ε, για δύο χώρε, παραδείγματο χάρη για την Ισπανία και τη Σουηδία, ότι θα έπαιρναν τα ίδια μέτρα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώ είναι οι διάφορε συνθήκε και οι διάφορε δομέ. Έτσι λοιπόν πρέπει να μείνουν αυτά στα χέρια των κρατών μελών, γιατί πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή σε ορισμένε περιπτώσει αφαιρεί ευελιξία από τα κρατημέλη, Δεν θα μακρηγορήσω εδώ, όμω ορισμένα παραδείγματα μπορούν να είναι παραδείγματο χάρη το άρθρο 13 με την ανάθεση καθηκόντων. Δηλαδή εδώ θεσπίζεται ένα σύστημα, όμως ε, δεν θέλουμε η Κομισιόν να νομοθετεί για κάθε καθήκον και επίσης νομίζουμε ότι πρέπει να επιτρέπεται περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη που ξέρουν καλύτερα τη δομή τους και την κατάσταση στο έδαφος τους και το σύστημα εγγραφής επίσης και ταυτοποίησης. Πρέπει επίσης στις βάσεις δεδομένων τα κράτη-μέλη να έχουν μία καλύτερη δυνατότητα διαχείρισης αυτών των βάσεων δεδομένων. Και εδώ επιμένω. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των ζώων σε ολόκληρη την Ένωση. Τη επικουρικότητα των κρατών μελών βρίσκεται στην ασφάλεια του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η Ισπανία πάντα αυτή τη θέση θα υπερασπίζει και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την προσέγγιση αυτή, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Εμείς τα κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσει μπορούμε να βελτιώσουμε τι κοινοτικέ αποφάσει. Για να μου επιτρέπετε και με αυτό θα κλείσω. Ε, εμείς ε, πιστεύουμε ότι σε ένα κανονισμό που μιλά για την υγεία των ζώων ε, λείπει αναφορά στα εργαστήρια αναφοράς, γιατί αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματο μας. Νομίζουμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να αναφερθούν αυτά τα ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς και να υπάρχουν και κάποιοι βασικοί κανόνες λειτουργίας. Νομίζουμε ότι είναι λοιπόν θεμελιώδε και μα λείπει στην πρόταση. Επίση θεωρούμε ότι πρέπει να εναρμονίσουμε περισσότερο και καλύτερα κάποια συστήματα ταυτοποίηση. Ξέρω ότι τη συζήτηση αυτή την έχουμε απευθεία με την Κομισιόν σε σχέση με τα άλογα, όμω ειλικρινά η σημερινή νομοθεσία που έχουμε για τα άλογα είναι εφιαλτική. Εμείς σας ζητάμε, σας παρακαλούμε να υπάρχει εναρμόνιση για να μπορεί να εφαρμοστεί με απλό τρόπο. Και τέλος, δεν θέλω να προσθέσω και κάτι που δεν υπάρχει στην παρουσίαση. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αποσαφινιστούν τα άρθρα 22 και 23 σε σχέση με τις επισκέψεις αξιολόγησης της υγείας των ζώων. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό όμως πρέπει να υπάρξουν κάποια στοιχεία αποσαφήνισης, να κατανοούμε σε τι αναφέρονται τα άρθρα αυτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε, μια, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Γέγκλε έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που ακούσαμε πένουσε για την έκθεση αυτή. Αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα στο δύσκολο αυτό θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Βόξχολμ. Ανέφερε ότι μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε μια, ένα νόμο περί υγείας των ζώων και μάλιστα θεωρεί ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό ε, νόμο που να ξεπερνάει δηλαδή τα εθνικά όρια. Ε, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα που έθεσε και ο Ισπανός ε, συνάδελφος. είναι δύσκολο το θέμα αυτό για μας. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό νόμο για την προστασία των ζώων, ποια ζώα θα πρέπει να καλύπτονται από έναν τέτοιο νόμο και υπό ποια μορφή. Μιλάμε μόνο για τα ζώα που καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα ή μιλάμε για όλα τα ζώα. Υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη ζώα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, θα πρέπει να διασαφινιστεί αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, κύριο Αλμάν Σαντελάρα. Σε πολλά μέρη της παρουσίασής σας αναφερθήκατε στα κράτη-μέλη, στα εθνικά κράτη. Επί της αρχής συμφωνούμε σε αυτό αλλά θα πρέπει να κάνουμε εδώ το διαχωρισμό. Τι θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη-μέλη και τι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ρυθμιστεί. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τρία θέματα όπου πιστεύετε ότι θα πρέπει η ρύθμιση να είναι ευρωπαϊκή, διότι το πρόβλημα ξεπερνάει τα, όρια, τα σύνορα των κρατών μελών. Και θα ήθελα να ε, θυμίσω σε όλους σας ότι έχουμε τώρα ένα νέο σύστημα προϋπολογισμού, το οποίο από τώρα θα αρχίσει να ισχύει. Εάν ε, λοιπόν έχουμε μια κρίση στον, ε, ε, στην τροφική αλυσίδα που να ξεκινά από ένα κράτος μέλος και να έχει επιπτώσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να στοιχίσει τελικά πολλά χρήματα η καταπολέμηση του προβλήματος αυτού. Εάν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση από ό,τι υπάρχουν στον προϋπολογισμό, οι γεωργοί θα πρέπει να καλύψουν το επιπλέον κόστος. Και αυτό θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κέκλε. Δίνω το λόγο στον κύριο Άγνιο. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια τον όσον είπε η Σπενίδα συνάδελφος, όσον αφορά την γκρίζα ζώνη, μας μίλησε και για μια λυπή μετάφραση κάποιου όρου στα ισπανικά. Εδώ προσοχή γιατί μπορεί να μπερδευτούμε. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ζώων. Οι δύο είναι εύκολο να οριστούν. Τα κατοικίδια και τα ε, ζώα για εκμετάλλευση στις εκτροφές. Μετά έχουμε τα αγρία ζώα, αλεπούδες, ασβούς κλπ. Ξέρουμε που ζουν. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία, μια τέταρτη κατηγορία, που είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί. Είναι τα κατοικίδια ζώα τα οποία δραπετεύουν, διαφεύγουν και παρέρχονται σε μια ελεύθερη κατάσταση. Σκύλοι για παράδειγμα. Και έχουμε και τα παράλληλα είδη, τα οποία ζουν και ελεύθερα, αλλά και σε αναπαραγωγή, όπως ο σολμός, όπως τα ελάφια και ούτω καθεξής. Ή τα άλογα, πόνοι στη χώρα μου υπάρχουν. Προσοχή λοιπόν στον ορισμό όλων αυτών των κατηγοριών ζώων. Ελπίζω να καταγράφει και η άποψή μου. Το άλλο θέμα είναι τα αντιβιωτικά. Ευχαριστώ που αναφέρατε την μεγάλη μείωση της χρησιμοποίησης, της χρήσης αντιβιωτικών. Πολύ και στην δική μου εκλογική περιφέρεια διαμαρτύρονται και λένε ότι οι κτηνοτρόφοι τρέφουν τα ζώα τους με αντιβιωτικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Χρειάζεται συνταγή καταρχήν για να χρησιμοποιήσει κάποιο αντιβιωτικά. Και ο γιατρός, ο κτηνίατρος πρέπει να πιστεί περί της αναγκαιότητας χρήσης του αντιβιωτικού. Εγώ Είμαι στον ε, τομέα και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν και περιορισμοί ακόμα και όσον αφορά την προληπτική χρήση αυτών των ε, αντιβιωτικών. Οπότε θα ήθελα αυτό το θέμα να κλείσει γιατί δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν ε, έχουμε άλλους που να έχουν ζητήσει το λόγο. Θα παρακαλούσα λοιπόν ε, τον καθηγητή Βόξχολμ να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση αφορούσε την νομοθεσία περί υγείας των ζώων. Τι εννοούσα. Στο πρόσχεσμα μέλλον ελπίζω θα θεσπιστεί και νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Το αν θα είναι κοινοτική νομοθεσία, εξαρτάται, είναι επιχείρημα υπέρ αυτού, είναι ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία δηλαδή, των ζώων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε λοιπόν μια παρανόηση και ζητώ συγγνώμη, είπα υγεία των ζώων, αλλά εννοούσα την προστασία των ζώων, συνθήκη ζωή, κλπ. Τώρα ω προς τα αντιβιωτικά. Χαίρομαι που ο βουλευτής από τον Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε το θέμα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να διαβάσουμε μακριά, δεν βλέπω το όνομά σας. Συμφωνώ όμως απολύτως. Έχουμε πάει μπροστά και εσείς λέτε ότι χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος. Βεβαίω. Αυτό μας απασχολεί και εμάς. Η νομοθεσία που συζητούμε θεωρώ ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε παρόμοιες επιτυχίες στο μέλλον, σαν αυτές που ζήσαμε στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν πετυχημένα παραδείγματα. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο των επιτυχιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι πολύ καλή πρόεδρος. Ο κύριος Αλμάν Σαντελάρα έχει το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξή. Αναφερθήκατε στο καθεστώς των κρατών μελών. Είναι ένα από τα πολύ δύσκολα πολύπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε κάποια πράγματα να γίνονται με τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της Ευρώπης, ενώ συμφωνούμε ότι υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία εντός της Ευρώπης όσον αφορά τη φύση, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις ε, κλπ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να πετύχουμε στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο εάν δεν έχουν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες τη δυνατότητα να προσαρμοστούν. Αυτό όμως είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Ε, Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Γιάγκλα. Να πω καταρχήν ότι εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος για την αναγκαιότητα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η νομοθεσία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες λειτουργίας, διαφορετικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε γιατί η υγεία των ζώων δεν έχει σύνορα και θέλω αυτό να ξεκαθαριστεί για όλους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ε, αυτοί οι κανόνες πρέπει να είναι τόσο αυστηροί που να φτάσουμε στο σημείο να ρυθμίζουν ε, και το τελευταίο κόμμα. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα όσοι είναι εκεί επιτόπου να έχει ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευελιξία και δυνατότητα να αλλάξει κάποιες αποφάσεις γιατί αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της κοινωτική νομοθεσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά τη νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε σε αυτή. Αλλά πρέπει να δώσουμε ευελιξία στα κράτη-μέλη για τα τελευταία στοιχεία. Διαφορετικά θα συναντήσουμε προβλήματα και έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα αυτό. Δεν ε, μιλάμε για κάτι καινούριο. Σε αυτή τη δύσκολη ισορροπία προσπαθούμε να συμβιώσουμε πάρα πολλά χρόνια και πάντοτε τα έχουμε καταφέρει επιτυχώ και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δύσκολη ισορροπία. Η κυρία Γιάννη με ρώτησε κάτι και θα σας ε, αναφέρω κάποια παραδείγματα. Έχουμε την ανάθεση καθηκόντων. Παραδείγματο χάρη, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει στην κοινωτική νομοθεσία ουσιαστικά ένας κατάλογος που καθορίζει πώς πρέπει να αντιθέτουν τα καθήκοντα, όμω, το κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει για την εκτέλεση των καθήκοντων, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει μια εκτελεστική πράξη κάθε φορά από την Κομισιόν. Τώρα, κινήσεις ε, εντός ε, των κρατών μελών, το ίδιο το εκτιμώντας αναγνωρίζει ότι το σύστημα ήδη λειτουργεί καλά. Γιατί να το αλλάξουμε. Και ένα ακόμη παράδειγμα, τρίτο παράδειγμα, είναι η νόση εκούσιας εξάλληψης. Δηλαδή, αν πρόκειται για ένα χαρακτήριο εκούσιο, πρέπει να υπάρχει ευελιξία για τα κρατημέλη. Πάντοτε λειτουργούσαν έτσι τα πράγματα στον τομέα αυτό και λειτουργούσαν καλά. Δεν είναι καινούριο λοιπόν να έχει ένα κρατός μέλος μία νόση και όλοι να την πληρώνουμε. Μπορώ να σα φέρω πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Εγώ ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τροποποιήσει την ε, χρηματοδοτική πρόταση ε, και θα προχωρήσει ανάλογα και με την ε, νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και σε σχέση με το θέμα των άγριων ζώων ή των ε, κόστων ζώων και αυτό είναι σημαντικό γιατί πρέπει και οι δύο αυτές κατηγορίες να είναι τμήμα της πρότασης. Βέβαια, τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μία κατηγορία και για την άλλη κατηγορία είναι διαφορετικά. Όμως και αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται γιατί έχουμε παραδείγματο χάρη και τα άγρια ζώα τα οποία επιδρούν με κάποια άλλα ζώα που είναι ελεύθερα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή βέβαια. Είναι διαφορετικά τα μέτρα ελέγχου γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε τα ίδια μέτρα για μια αγελάδα και για ένα άγριο ζώο. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσει σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βόξχολμ και τον κύριο Αλμάνσα για τις παρουσιάσεις τους. Και περνάμε σε δύο άλλους εμπειρογνώμονες. Έχουμε τον κύριο Γιάν Παραντότα που είναι Διευθυντής ε, του Τμήματος ε, Τροφικής Ασφάλειας ε, και Εκτινιατρικών Θεμάτων στην Πολωνία. Καλώς ήρθατε. Και έχουμε και την κυρία Λουίζα Πέιξε. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο, στην Πορτογαλία. Και είναι και μέλος ε, της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΦΣΑ για τους βιολογικούς κινδύνους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Δίνω πρώτα τον λόγο στον δόκτωρο Αμπραντότα. Δέκα λεπτά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Na samym początku chciałem serdecznie podziękować za. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην συζήτηση σήμερα. Αποτελεί χαρά για μένα γιατί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια Εργάζομαι ως ε, υπεύθυνο κτηνιατρικών θεμάτων στην ε, αντιπροσωπεία της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πράγματα λοιπόν από την πολωνική οπτική γωνία. Αλλά και δύο λόγια για την τρέχουσα κατάσταση ενώψη και της ε, προτινόμενη νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Έχω κάποιο σχέδιο Παρ' όλα αυτά επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε δύο-τρία σημαντικά θέματα. Τα πιο σημαντικά, γιατί το γενικό μέρο νομίζω καλύφθηκε από του προλέλησεντες. Συμφωνώ με τα όσα ήδη ακούστηκαν εν γέννη. Θέλω να υπογραμμίσω όμως ότι η νέα προσέγγιση είναι πραγματικά νέα. Όχι μόνο για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς. Φαίνεται ότι είμαστε έτοιμοι να θεσπίσουμε κανόνες οι οποίοι δεν συνάδουν πάντοτε με τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών. Το θέμα είναι εμείς να ενερμονίσουμε τους κανόνες μας. Με τους ε, αρμοδίους οργανισμούς παγκοσμίω για την υγεία των ζώων και με άλλους οργανισμούς. Ο βασικός στόχος ήταν, επαναλαμβάνω, να απλουστεύσουμε και να νερομονήσουμε τους δικούς μας κανόνες, τους φυστάμενους κανόνες. Θελήσαμε επίσης να γίνουμε καλύτεροι στην αντιμετώπιση των κρίσεων να μπορούμε να επεμβαίνουμε εγκαίρως, το συντομότερο δηλαδή δυνατόν, στην περίπτωση κρούσματος κάποιας μολυσματικής ασθένειας και δι ασθένειας, ε, ζωνός που θα μπορούσε να προσβάλλει και τους ανθρώπους. Το σημαντικότερο στοιχείο της πρότασης είναι η κοινή ευθύνη. Όχι μόνο των ευρωπαϊκών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την υγεία των ζώων, αλλά και άλλων φορέων και όλων των εμπλεκομένων των ιδιοκτητών των ζώων ενώσεων, παραγωγών, εκτροφέων κλπ. Χρειάζεται συνεργασία. Αυτή η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί. Διότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι μολυσματικές, οι μεταδιδόμενες ε, ασθένειες, ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα. Ένα από τα δύνατα σημεία της πρότασης, το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, αλλά θέλω να σταθώ λίγο εδώ. Ένα λοιπόν από τα δύνατα σημεία είναι η γενικότητα της νομοθεσίας. Φυσικά δεν είναι εύκολο να πλουστεύεις αφενός και να κωδικοποιείς αφετέρου. Όμως, κάποιες ειδικότερε προσεγγίσεις πιστεύω θα ήταν ευπρόσδεκτες. Σε ορισμένες διατάξεις βλέπω γίνεται αναφορά σε άλλους κανόνες πράγμα το οποίο καθιστά την πρόταση δυσνόητη. Ως προς τα θετικά, θα έλεγα ότι πρώτον, η πρόταση εξασφαλίζει περισσότερη ευελιξία, ανάλογα με την νόσο. Επιπλέον, επιτρέπει νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση ζωών νόσων, ασθενειών γενικότερα και διζωνώσεων και εστιάζεται στην πρόληψη παρά τη θεραπεία. Επίσης, η πρόταση θέτει μια νέα προσέγγιση στο θέμα του εμβολιασμού με τον οποίο βεβαίως έχουμε αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες. Χάρη στον εμβολιασμό, για παράδειγμα, δύο χρόνια πριν, κήρυξαμε ως ολοκληρωμένη την εκρίζωση μιας από τις πιο σημαντικές ασθένειες των βοηδών. Όπως έχουμε κάνει και με μερικέ ασθένειες τους ανθρώπους. Επειδή τώρα κάποιο αναφέρθηκε στην Λίσα, ο βουλευτή από το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα ανέφερε την απειλή από την Λίσα. Δυστυχώ είναι πολύ επικίνδυνη όσο, όντω, η οποία ως τώρα είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς σε όλη την Ευρώπη και στην Πολωνία. Στην Πολωνία γίνονται τώρα εμβολιασμοί στα σύνορα με την Ουκρανία, στις περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, για να μην περάσει η ασθενεία στη χώρα μας. Σκέφτομαι όμως ε, όχι μόνο εμάς, αλλά και τους γειτονές μας. Πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε και τις γειτονικές μας τις όμορες χώρες στο παιχνίδι. Μία από τις πτυχές της πρότασης αφορά κάποιες νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία και συνάρτηση με την κοινή ελευθερική πολιτική, την κοινή, την κοινή αγροτική πολιτική κλπ. Για να κλείσω αυτήν την σύντομη εισήγηση, επιτρέψτε μου να πω ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα Οι κανόνες και οι αρχές που προβλέπουμε το σχετικό σχέδιο θα περιορίσουν ακόμη περισσότερο κάποιες από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες. Μην ξεχνάτε την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, η οποία μπορεί να προήλθε από τον νότο της Αφρικής, αλλά μην ξεχνάτε και την Ανατολική Αφρική. Όπως επίσης και από την Ανατολική Ευρώπη, μόλις 160 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Η απόσταση είναι μικρή. Θα μπορούσε η εξαπλωσή της στη χώρα μας να επηρεάσει πάρα πολύ την κτηνοτροφία. Εν γέννη λοιπόν, η έννοια της προστασίας των ζώων με τρόπο γενικό δεν είναι η καλύτερη λύση. Διότι υφίστερε βεβαίω ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να επαναλάβουμε να επικαλυφθούμε με υφισταμένη νομοθεσία. Αυτά ως προς την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα την καθηγήτρια Πέιξε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Many thanks for the invitation. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Πόλσεν. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να μιλήσω για την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, γιατί είναι ένα θέμα που περιλαμβάνεται και σε αυτή την νομοθετική πρόταση και χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται το θέμα αυτό, γιατί ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες εργαζόμαστε στο θέμα της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά, όχι μόνο στα ζώα, αλλά και στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Μέσα σε λίγες διαφάνειες ε, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποιες πληροφορίες που θεωρώ σημαντικές για την κατανόηση του προβλήματος και θα μπορούσα να προτείνω νομοθετικά μέτρα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτό το, να περιορίσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Έχουμε αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται για τους ανθρώπους και τα ζώα πάνω από 50 χρόνια και τα περισσότερα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται σε ζώα για παραγωγή τροφίμων είναι ταυτόσιμοι ενικούν στην ίδια κατηγορία με τα αντιβιωτικά για τους ανθρώπους. Αν μπορείτε να δείτε εδώ στη διαφάνεια, μόνο τα αντιβιωτικά με μαύρα γράμματα είναι αυτά που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ζώα που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων από τα τέλη της δεκαετίας του 70 τουλάχιστον ε, τα αντιβιωτικά που εισήχθησαν στην αγορά, εισήχθησαν νέα αντιβιωτικά μάλλον στην αγορά ε, επειδή είχαν εμφανιστεί ήδη φαινόμενα ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά και φτάνουμε τώρα στην ε, τελευταία περίπτωση που δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε νόσους στον άνθρωπο με τα αντιβιωτικά. Έχουμε εδώ λοιπόν ε, δύο κατηγορίες ε, όπου χρησιμοποιούνται περισσότερα αντιβιωτικά. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το 50% των αντιβιωτικών και πάνω χρησιμοποιούνται στα ζώα. Και η συνέπεια είναι ότι και ε, οι άνθρωποι και τα ζώα ευθύνονται για αυτή την ευρεία διάδοση των βακτηρίων. Φυσικά, προκειμένου να καταλάβουμε την πλήρη εικόνα, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι αντιβιωτικές πολιτικές ποικίλουν. Ανάλογα με τη χώρα, ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες στον κόσμο χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά για οτιδήποτε και η έλλειψη ελέγχου ή ρύθμισης αποτελεί πραγματικότητα στις περισσότερες χώρες του κόσμου, κυρίως όπου έχουμε τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Επίσης υπάρχουν και σωρευτικά σορευτικές συνέπειες, σωρευτικές παρενέργειες, ε, σημαντικό και αυτό στοιχείο του προβλήματος να σας επενθυμίσω ότι οποιαδήποτε χρήση αντιβιωτικών, είτε είναι κατά είτε όχι, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κάποια στελέχη ανθεκτικότητας και αυτά οδηγούν σε μετάλλαξη των γονιδίων ε, ή σε πρόσληψη γονιδίων. Ή σε πρόσκτηση γονιδίων. Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρξουν δυνατότητες ανθεκτικότητας ε, στα αντιβιωτικά και ξέρουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για οποιοδήποτε ε, θέμα ε, ανθεκτικότητας ε, θα πρέπει να δούμε ότι γίνεται μία διάδοση μέσω των γονιδίων μεταξύ των ε, ειδών και των γενών. Και γίνεται αυτό με σύζευξη, μετασχηματισμό και μεταγωγή. Αλλά επίσης ε, πρέπει να δούμε και τι γίνεται στην ε, συνεπιλογή. Γιατί πρέπει το ε, ξέρουμε σήμερα ότι τα αντιβιωτικά μπορεί να μιλήσουν το πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι η ανθεκτικότητα στα γονιδία μπορεί ε, να ε, μας ε, οδηγήσει στην ενεργοποίηση ορισμένων βακτηρίων και αυτή η συσσόρευση της ανθεκτικότητας στο ίδιο γονίδιο θα ευνοήσει την συνεπιλογή και αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ένα γονίδιο σε μία πλατφόρμα αυτό θα αντιστέκεται σε οποιοδήποτε αντιβιωτικό χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, είτε χρησιμοποιήσω το αντιβιωτικό 1 είτε το αντιβιωτικό 2, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, αν ε, δεν ξέρουμε πραγματικά τι κάνουμε. Τώρα επανέρχομαι σε αυτή τη διαφάνεια για να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα δύο hot spot ανθεκτικότητες είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή τα ζώα και οι άνθρωποι. Και σε ό,τι αφορά τα ζώα πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε πολλά στοιχεία που μας δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατηγορία σε ό,τι αφορά τα βακτήρια, το οίκο, e. όλοι ε, και άλλα βακτήρια που θεωρούμε ότι έχουν ήδη εκριζωθεί. Και στην περίπτωση αυτή βλέπετε ότι υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητα σε πολλά αντιβιωτικά υπάρχουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σαλμονέλα ε, και υπάρχει και ανθεκτικότητα σε δύο ομάδες αντιβιωτικών αρκετά σημαντικών που τα βλέπετε με κόκκινο περίγραμμα. Όχι μόνο στη Σεφοταξίμ ε, αλλά και στην Αμπικιλίνη και ξέρετε ότι ε, για την περίπτωση του Σύπροφλο Ξασίν έχουμε μεγάλο βαθμό ανθεκτικότητας στη σαλμονέλα όπου χρησιμοποιείται αυτό το αντιβιωτικό. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ε, να υπάρχει χρήση αυτού του αντιβιωτικού ε, που στην περίπτωση που χρησιμοποιείται έχουμε ανθεκτικότητα στη σελμονέλα. Εδώ βλέπετε λοιπόν κάποια στοιχεία της ΕΦΣΑ. Βλέπετε εδώ για το ότι τη Εδώ για να κατεπολεμηθεί αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον πέντε σημαντικά αντιβιωτικά και ορισμένες ε, χώρες έχουν αναφέρει ανθεκτικότητα στα ε, σεφαλοσπρίν. Άλλο παράδειγμα αφορά το καμπυλοβακτήρια. Έχουμε ε, τη πιο συχνή γυζονόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα καμπυλοβακτήρια βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται και στα πουλερικά, αλλά βλέπετε και υψηλά ποσοστά σε άλλα ζώα. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τα στοιχεία από τις κάτω χώρες. Συλλέγονται στοιχεία από το 92 σε σχέση με τα καμπυλοβακτήρια και τα στοιχεία ανθεκτικότητας ε, στα αντιβιωτικά αφορούν το σιπλοκροφετσίν, το ritromycin και άλλο ένα αντιβιωτικό και να σας πω ότι το ritromycin και το σιπλοφαξίν είναι τα αντιβιωτικά που, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καμπυλοβακτηρίωσης και βλέπετε ότι υπάρχει αυξητική τάση ανθεκτικότητας ε, στα αντιβιωτικά και αυτό αντικατοπτρίζει τι έχει γίνει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, ε, βλέπουμε ότι ε, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία μας επιτρέπουν να έχουμε σαφέστερη εικόνα του προβλήματος. Μερικές φορές ε, βέβαια υπάρχουν και αλλαγές και σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ένα αυξημένο αριθμό των μολυσματικών ασθενειών ε, και του χαρακτήρα αυτών των νόσων στην Ευρώπη. 25.000 ήταν το χρόνο σχετίζονται με αυτό το πρόβλημα και επίση έχουμε και αύξηση ε, του θανάτου και του κόστους βέβαια. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την επιτακτική ανάγκη της, ε, του φαινομένου της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά. Πάντως, ε, η χρήση των αντιβιωτικών θεωρείται ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας ε, στα βακτήρια, των βακτηρίων. Ε, μία πτυχή βέβαια είναι και η παγκοσμιοποίηση στο εμπόριο των ζώων ε, και στην παραγωγή τροφίμων. Αυτά από μένα και αν έχετε ερωτήσεις ευχαριστώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ε, θεωρεί ότι αυτό είναι ένα από, μία από τις τρεις ή τέσσερις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρωπότητα στο μέλλον. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Υπάρχει λοιπόν κανείς που να έχει ερωτήσεις, που να θέλει να θέσει. Μακίνες. Η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πολύ γρήγορη, αναλυτική και, ε, και αναλυτική η τελευταία παρουσίαση και θα ήθελα παρακαλώ ε, να μας την υποβάλλετε γραπτός. Ε, δεν βλέπω και πολύ καλά, δεν μπόρεσα να διαβάσω τις διαφάνειες. Ήταν πολύ αναλυτική και λεπτομερής και πλήρης η παρουσίασή σας. Είναι λοιπόν δυνατόν να μας ε, την υποβάλλετε σε χαρτί. Και μια και πήρα το λόγο, μιλήσατε για την χρήση των αντιβιωτικών, είναι πλοκό το θέμα. Εάν βρισκόσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα κάνατε όσον αφορά τις τρεις ε, προτεραιότητες ε, για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, ώστε να επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης των αντιβιωτικών όπου ενδείχνεται στη γεωργία και πώς ε, μπορούμε να καλύψουμε τις ανησυχίες που έχετε όσον αφορά την ανθεκτικότητα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, θα σας υποβάλω γραπτός ε, τις ε, διαφάνειες αυτές ε, και με παραπομπές που να στηρίζουν τις θέσεις μου. όσον αφορά το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κυρίως δύο πτυχές. Πρώτον, πώς μπορεί να μειωθεί η πώς μπορεί να, να ε, μειωθεί η απειλή βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να μειωθεί η χρήση των αντιβιωτικών. Θα πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά που έχουν εισαχθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά αυτά για μένα δεν θα αποτελούσαν προτεραιότητα. Ε, για μένα προτεραιότητα αποτελούν τα αντιβιωτικά τρίτης γενιάς. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στα αντιβιωτικά ε, για τα οποία η ανθεκτικότητα έχει εξαπλωθεί περισσότερο. Είναι σαφές ότι αν δεν μειωθεί και η χρήση των αντιβιωτικών, ε, μπορούμε στα ζώα, στους ανθρώπους, ε, διότι είναι κάτι που ισχύει για όλους, μπορεί να έχουμε ε, αυτά τα ανθεκτικά βακτήρια. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με την εμφάνιση της ανθεκτικότητας αλλά και την εξάπλωσή της. Θα πρέπει να μειώσουμε τις ε, λοιμώξεις. Ε, είναι λοιπόν ε, σημαντικό να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά την βιοασφάλεια και μπορούμε να επικεντρωθούμε στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι στα πουλερικά έχουμε τα καμιλοβακτήρια Υπάρχουν ενώσει καταναλωτών ε, που ε, δίνουν στοιχεία σχετικά με τον επιπολασμό ε, της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά των αντιβιωτικών τρίτης γενιάς στα πουλερικά. Αυτά τα προϊόντα πολλούνται σε αρκετές χώρες και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και ε, θα πρέπει... Όσον αφορά λοιπόν τις κεφαλοσπορίνες, ε, να ε, περιορίσουμε τις δυνατότητες πώληση ζώων που ήδη έχουν μολυνθεί με αυτά τα ανθεκτικά βακτήρια. Επίσης έχουμε και άλλες σημαντικές στοιχές. Μία από αυτές είναι να ξέρουμε πού βρίσκονται τα βασικά προβλήματα ε, για να μπορέσουμε να ε, περιορίσουμε την εξάπλωση. Ε, ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι είχαμε στη Γερμανία μια εμφάνιση σαλμονέλας ανθεκτική στα αντιβιωτικά, στα, στους χείρους και στα πουλερικά. όταν χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα που έχουμε για να αντιμετωπίζουμε την ανθεκτικότητα απέναντι σε πολλά φάρμακα, το MDR δηλαδή στους ε, ανθρώπους, δεν έχουμε πια άλλα μέσα στη διάθεσή μας. Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα να περιορίσουμε την εξάπλωση. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε το πρόβλημα να καθορίσουμε τα, τα σωστά μέτρα για να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες. Πρέπει να σκεφτούμε τους παραγωγούς που πρέπει να επιβιώσουν, πρέπει όμως να διαφυλάξουμε και την υγεία μας. Να αναφέρω και ένα άλλο δύσκολο θέμα, ε, και άλλο, ε, και άλλο ένα ε, σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της υγιεινής. Εάν βελτιώσουμε την υγιεινή, μειώνουμε την δυνατότητα εξάπλωσης των ανθεκτικών αυτών βακτηρίων. και έτσι αποχωρίζουμε το πρόβλημα αυτό από την ε, ε, ε, ζωική παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μας στείλετε τα έγγραφα, διότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συνάδελφοί μου να καταλάβουν σωστά τι ακριβώς συζητάμε εδώ. Έχουμε επιφανειακές γνώσεις, όχι όμως αρκετές ειδικέ γνώσεις στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά και τους δυο σας. Και έχουμε τώρα τους, τους δύο επόμενους ομιλητές. Θα προσπαθήσω να προφέρω σωστά τα ονόματα. Ε, Ελσανόφσκι, τον καθηγητή Ελσανόφσκι, ζητώ συγγνώμη λέει ομιλήτρια. Από ε, Ίδρυμα Κοινωνιολογίας από την ε, Πολωνική Ακαδημία ε, Ζω, Ζωολογίας, συγγνώμη, το Ινστιτούτο Ζωολογίας ε, στην Πολωνική Ακαδημία Επιστημών και τον κύριο Μαρίνο Κόντου που είναι διευθυντής της Περιφερειακής Ένωσης Αγροτών στη Σαρδινία, στην Ιταλία. Δίνω το λόγο πρώτα. στον κύριο Ελζανόφσκι. Ε, Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου τιμή που παρευρίσκομαι απόψε. Ο χρόνος βεβαίως πιέζει, οπότε περνάω κατευθείαν στα θέμα μου. Όπως ε, όλοι συνομολογούν, η πρόταση είναι υπερβολικά γενικόλογη. Συμφωνώ με όσους το τόνισαν. Ανησυχώ διότι είναι μάλλον υπερβολικά γενικόλογοι, όπως είπαμε, πολλές, υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις και μεγάλη διακριτική ευχαίρεια όσον αφορά την εφαρμογή. Ανησυχώ ως κάποιος που έχει πείρα με την εθνική μας νομοθεσία. Στην Πολωνία γνωρίζω πόσο καλά τα πηγαίνουν κάποιες χώρες μέλη και πώς άλλες καταφέρουν να ξεφεύγουν από το δίκτυο της νομοθεσίας. Αυτά ισχύουν παντού. Η Πολωνία δεν είναι εξαίρεση. Και αυτό είναι ακριβώς και το πρόβλημα με την κοινοτική εν γέννη νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα. Κάποιες χώρες έχουν μια μινιμαλιστική πολιτική, κάνουν το λιγότερο που μπορούν όσο πιο αργά μπορούν Κάποιες άλλες είναι πιο αποτελεσματικές. Ο νομοθέτης λοιπόν πρέπει αυτό να το γνωρίζει. Και θα σας δώσω παραδείγματα. Δεν θα σχολιάσω φυσικά το σύνολο της πρότασης. Τα παραδείγματά μου είναι εκ των πραγμάτων αποσπασματικά. Ενδέχεται να, φερούν, να φορούν κατά κύριο λόγο την Πολωνία. Πρώτη αδυναμία, πρώτο ελάττωμα. οι έλεγχοι επιβάλλονται μόνο σε μια κατηγορία και μόνο εκμεταλλεύσεων. Άρθρο 24 συγκεκριμένα, όπου ορίζεται η συχνότητα και ο τύπος επιχείρησης που υπόκειται σε επιθεωρήσεις από κτηνιάτρους εν προκειμένου για τους σκοπούς του ελέγχου της υγείας των Αυτό, αυτή η συχνότητα δεν καθορίζεται. Λόγω των γνωστών πιέσεων από τα κράτη-μέλη, η πρόβληψη αυτή, αυτή, μάλλον η έλλειψή της, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικότερες παραλήψεις στο σύστημα ελέγχων. Γι' αυτόν τον λόγο, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω το ψήφισμα της συνέλευσης των Πολωνών κτηνιάτρων. Είναι κάτι σαν ένα κτηνιατρικό επιμελητήριο, αν θέλετε. Με το οποίο οι κτηνίατροι, οι Πολωνοί κτηνίατροι, εκφράζουν την πεποίθηση ότι πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη συχνότητα έξι μηνών στις παραγωγικές εκμεταλλεύσεις, στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και να μην αφήνεται αυτό στη διακριτική ευχέρεια των κρατομέλων. Τουλάχιστον λοιπόν εξαμηνιαίες επιθεωρήσεις. Το άλλο ζήτημα, εξίσου σημαντικό με την συχνότητα των επιθεωρήσεων και την υποχρέωση διενεργίας κτηνοτροφικών ε, ελέγχων, είναι το θέμα των πιστοποιητικών. Άρθρο 140 της ε, πρότασης. Η πρόταση απαιτεί πιστοποιητικό εντός του κρατούς μέλους. Ξεχνούμε εδώ τις μεταφορές μεταξύ κρατών μελών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και μόνο στη μεταφορά εντός κρατούς μέλους θα περίτε μόνον εφόσον τα ζώα μεταφερθούν από περιοχές που τελούν υπό περιοριστικά μέτρα. Αυτές είναι περιοχές με κρούσματα, για παράδειγμα, κάποιες κίνδυνης ασθένειας. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ρύθμιση συνεπάγεται του κινδύνου εξάπλωση ασθενειών σε τοπικό επίπεδο. Τα ζώα θα κυκλοφορούν ελεύθερα από αγορά σε αγορά. Δείτε τι έγινε με, την... με τον Αφθόδη πυρετό το 2001 στην Μεγάλη Βρετανία. Ξέρουμε πολύ καλά πως ε, η ασθενή εξαπλώθηκε στην αγορά. Λοιπόν, οι Πολωνοί κτηνίατροι πιστεύουν ότι το πιστοποιητικό υγείας πρέπει να πετείται για κάθε μεταφορά ζώων και όχι μόνο στις προαναφερθήσεις περιπτώσεις, στις ειδικέ δηλαδή περιπτώσεις ε, που έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα σε συγκεκριμένη περιοχή. Οι ανταλλαγές, οι αγροπολισίες ε, ζώων είναι ο τρόπος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Αυτό ισχύει και για την Πολωνία αλλά και αλλού. Πέρσι 100.000 ζώα διακινήθηκαν σε 50 αγορές στην Πολωνία, νομίμως και παρανόμως. Σύμφωνα με ΜΚΟ, δύο ΜΚΟ, μια γερμανική και μια πολωνική, που ασχολήθηκαν με το θέμα στην Πολωνία. Ακόμη και στις νόμιμες αγορές, εκεί όπου υπάρχουν κτηνίατροι που δημιουργούν ελέγχους κλπ. Σε αυτές τις αγορές διακινούνται άρρωστα οι νεκρά ζώα. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι τελευταίες επιθεωρήσεις από το FVO, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δυστυχώς αυτή η ιστορία συνεχίζεται ανεμπόδιστα. Κανείς δεν αντέδρασε, κανείς δεν έκανε κάτι μετά από την δημοσίευση της επικριτικής έκθεσης του FEO για την Πολωνία. Η ιστορία αυτή παραλαμβάνω συνεχίζεται και από ό,τι ξέρω όσον αφορά τους κτηνεδρικούς ελέγχους η ιστορία αυτή θα συνεχιστεί όσο η παράνομη διακίνηση στην Πολωνία αξιοποιεί τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δείτε τις φωτογραφίες αυτές που λήφθησαν Ιούλιο παρακαλώ του 2013. Αυτές οι πρακτικές σημαίνουν ότι άρρωστα είναι κραζό μεταφέροντας στα σφαγεία. Στην Πολωνία ξέσπασε ένα σκάνδαλο τον Μάρτιο του 2013 όταν συνειδητοποίησαμε την κατάσταση Στη συνέχεια ο διευθυντής της ε, διεύθυνση κτηνιατρικής είπε ότι περνάμε σε ένα καθεστώ μηδενική ενοχή και κάτι έγινε. Ε, η βελτίωση ήταν όμω μερική και μόνο. Τέτοιου είδου ε, διακινήσεις ζώων γίνονται ακόμη και σήμερα σε διάφορε αγορέ στην Πολωνία. Ούτω ή άλλω αυτά που σα δείχνω έγιναν μόλι τον περασμένο Ιούλιο. Αυτό το οποίο κάνει το πρόβλημα ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι ορισμένε τέτοιε αγορέ είναι επίσημε. Υπόκειται σε ελέγχου. Κάποιε όμω είναι εντελώ παράνομε. Δεν γίνονται δηλαδή καν κτηνιατρικοί έλεγχοι. Οι κτηνίατροι μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις αρνούνται να διενεργήσουν ελέγχους το οποίο είναι εντελώ παράλογο για μένα. Είναι σαν ε, ένα εγκληματία να πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να τελείπω τον έλεγχο της αστυνομία. Τα λέω όλα αυτά και σας δείχνω ότι σα δείχνω αυτές τις ε, τρομακτικές φωτογραφίες διότι έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι αυτές οι αγορέ δεν είναι μόνο πολωνικό πρόβλημα ούτε, μόνο στην... ούτε υπάρχουν μόνο στην Ανατολική Ευρώπη είναι θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ζώων αλλά και την υγεία των ζώων όπως υπογραμμίζεται από την υπόθεση του αυθόδου σπιριτού στην Μεγάλη Βρετανία. Συνεπώς, δεν βλέπω γιατί αυτή η πρόταση θεωρείται λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Θεωρώ ότι η πρόταση λοιπόν δεν βαίνει προς επίλυση των ζητημάτων. Χρειαζόμαστε πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία για να πειθαρχήσουμε κάποιες αρμόδιες αρχές, οι οποίες όπως στην περίπτωση της Πολωνίας ανέχονται την παραβίαση το, της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων και την προστασία των ζώων. Τέλος, Θα συμφωνήσω με την κυρία Πόλσεν και την έκθεσή της ως προς το ότι δεν υπάρχουν διατάξεις για να μειωθεί η μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων διαπιστώνει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την διάδοση ασθενειών στην Ευρώπη. Απελούνται μολύνσεις διότι τα ζώα μπορούν να μολύνουν το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της μεταφράσης ή κατά την αφήξή τους. Σε πολλές περιπτώσεις της σαλμονέλωσης αυξάνει έτσι και ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Θεωρώ ότι ο προτινόμενος κανονισμός θα έπρεπε τουλάχιστον να παίρνει προς την κατεύθυνση της μείωσης του όγκου και της διάρκειας της ζών των ζώων και τέλος επειδή ο χρόνος μου τελειώνει, θα ήθελα να πω ότι στις μεγάλες εκτροφές ε, το θέμα της προστασίας και της υγείας επικαλύπτεται. Τα δύο αυτά θέματα είναι αλληλένδετα. Το να τα ξεχωρίσουμε για λόγους κανονιστικούς θα έχει αρνητικές και μόνο επιπτώσεις και στους δύο τομείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες που μας δείξατε. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Δίνω τώρα τον λόγο στον Μαρίνο Κόντου, που ε, είναι επικεφαλής της Ένωσης Γεωργών στη Σαρτενία. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας για την πρόσκληση. Για μένα είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι εδώ σήμερα και να φέρω στο Κοινοβούλιο την φωνή των εκτροφέων. Είμαι ο Μαρινό Κόντου ε, και είμαι διευθυντής ε, της Περιφερειακής Ένωση Κοινοτρόφων της ε, Σαρδινίας και υπάρχουν και κάποιες διαφάνειες. Εκεί θα δείτε μια παρουσίαση του Άρας, δηλαδή τη υπηρεσίας που προσφέρουμε εμεί σε όλους τους κτηνοτρόφους. Είμαστε ε, μια ένωση ιδιωτικού δικαίου και έχουμε τέσσερις εταίρους και λειτουργούμε στα πλαίσια της πολιτικής που διέπεται από την Κτηνοτροφική Ένωση της Ιταλίας. Στην ε, Σαρδινία εμείς διαχειριζόμαστε το επιχειρησιακό σχέδιο ε, τεχνικής βοήθειας ε, και αποτελούμαστε από μία, βοηθούμαστε μάλλον από μία δομή 230 τεχνικών γεωπόνων και κτηνιάτρων που καθημερινά ενημερώνουν και βοηθούν τους κτηνοτρόφους για τις θεματικές του τομέα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι γνωρίζουμε ε, τα προβλήματα της ζωοτεχνίας. Η προσέγγιση είναι διατομεακή, είναι πολυτομεακή, βασίζεται στην πρόληψη, χρησιμοποιώντας τα μέσα που προσφέρονται από τις περιφερειακές πολιτικές. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι οι στόχοι που επιδιώκει η Κομισιόν ε, για την αναθεώρηση της σημερινής νομοθεσίας στο θέμα της υγείας των φυτών και των ζώων και του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού ε, και των επίσημων ελέγχων μας βρίσκουν γενικά σύμφωνους. Η πρόθεση όλων των πρωτοβουλειών για την εγγύηση της ε, προστασίας και της υγείας των ζώων έχει ωφέλη στο ζωοτεχνικό τομέα και ταυτόχρονα προωθεί την εφαρμογή των βελτιστικών πρακτικών. Επίσης, συμφωνούμε στο ότι στο να υπάρχουν καλές συνθήκες υγείας των ζώων είναι μια προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη και για να εγγυηθούμε το κατάλληλη ποιότητα των τροφίμων στον καταναλωτή. Ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν οι κτηνοτρόφοι ε, για την προστασία της υγείας των ζώων πρέπει να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί. Οι κτηνοτρόφοι είναι η πρώτη γραμμή εποπτείας ε, και ουσιαστικά προστατεύουν τα ζώα και καθιστούν αδιαχώριστο το διώνυμο ευημερία και αηφορία. Ο ε, θα πρέπει οι εκτροφείς να εμπλέκονται πλήρων σε οποιοδήποτε σχεδιασμό για την υγεία ε, των ζώων και να, θα πρέπει να συνεισφέρουν οι κτηνοτρόφοι στην επίτευξη των στόχων για την αποτελεσματική εφαρμογή του πακέτου που προτείνεται. Είμαστε πεπισμένοι για την συνεργική συνεργασία όλων ε, των ε, εμπλεκομένων, όμως ε, θέλουμε να προβλέπετε όχι η ποινικοποίηση, αλλά η χορήγηση κινήτρων ε, θα θέλαμε να υπάρχει προσχώρηση στο σύστημα των λειτουργικών ελέγχων που θα μπορούσαν να αποτελούν ένα πρώτο σύστημα παρακολούθησης του κινδύνου και σημαντική συνιστόσα ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης των επιδημιών. Μέσω κάποιων σχεδίων χορήγησης συμβουλών θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να ενημερώνονται ε, και θα πρέπει να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους ως μια ομάδα που παράγει τρόφιμα για τους υπόλοιπους πολίτες, τους καταναλωτές. Με την πλήρη εμπλοκή των κτηνοτρόφων θα μπορούσε να δημιουργηθούν οι συνθήκε για μια αποτελεσματική πρόληψη των ζωνώσεων. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή όπου υπάρχουν ε, πραγματικά κάποιε ντροπιαστικέ ζωνώσει, αλλά υπάρχουν και κάποια ενάρετα σχέδια, όπω ε, παραδείγματο χάρη η προστασία των εγωπροβάτων, όπου ο κτηνοτρόφο συμμετέχει ε, και ενημερώνεται στις διαδικασίες βελτίωσης της προστασίας ε, των κοπαδιών. Και αυτό έχει επιτρέψει να παράξουμε ε, τυρί ε, από γάλα, από εγωπρόβατα εξαιρετικής ποιότητας. Και το 65% του γάλακτος στην Σαρδινία ε, μπορεί να μας ε, οδηγήσει στην παραγωγή τυριών ακατέργαστου, του γάλακτος. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε ότι πάντοτε μιλάμε για τα σκάνδαλα και όχι για τα θετικά. Όμως θα πρέπει με τους κτηνοτρόφους να συνομιλούμε και όχι να χρησιμοποιούμε τη διαδικασίες. Η οργάνωση των κτηνοτρόφων πάντοτε θα εργαστεί στο πλάι των κτηνοτρόφων σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα. Οι δικοί μας γεωργοί και κτηνοτρόφοι πρέπει να προστατεύονται γιατί παράγουν τροφή που όλοι εμείς οι πολίτες καταναλώνουμε. Γι' αυτό στρέφουμε στους πολιτικού, χρειαζόμαστε και τη δική σας υποστήριξη. Πράγματι με την παγκοσμιοποίηση δημοκρατία γίνεται ένα πολιτικό εργαλείο των πολυεθνικών που προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν για το δικό τους συμφέρον. Η πολιτική ε, θα ε, έπρεπε ε, να ωφελεί όποιον καλλιεργεί τη γη εσείς και εμείς ε, θα πρέπει να είμαστε αυτοί που προστατεύουν ε, καλύτερα τη βιοπικιλότητά μας ε, και τους παραγωγούς μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία με τη φύση για να έχουμε μια βιώσιμη εφορία για τις επόμενες γενιές. Και έχουμε το παράδειγμα της Αρδινίας αυτές τις μέρες δυστυχώς ε, και βλέπουμε τι έχει γίνει με τους κατακλυσμούς όπου ο άνθρωπος δεν σέβεται τη φύση και χτίζει ε, πάνω σε ποτάμια και σε ρήματα προκύπτουν θάνατοι. Εμείς η ε, Ιταλία αναγνωριζόμαστε στον κόσμο επειδή έχουμε ένα μεγάλο ταλέντο που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει δηλαδή αναζητούμε μανιωδώς την ποιότητα και έχουμε και το θέμα της ε, συνήθειας. Ε, αυτό μας ξεχωρίζει στη δουλειά που κάνουμε. Η ίδια έννοια θα πρέπει να εφαρμοστεί και για την ποιότητα της τροφής σε σχέση με το πώς παράγεται, πώς καλλιεργείται, πώς, ε, είναι, πώς γίνεται η επεξεργασία και πώς μαγειρεύεται. Αυτές ε, τις έννοιες θα πρέπει να προστατεύσουμε. Κάθε παραχώρηση ε, που γίνεται σε όσους θέλουν να εξελίψουν τα πάντα είναι ένα βήμα προς ε, την παραγκόνηση του τομέα και κάθε σημείο που κατακτώμε σημαίνει ότι εγγυόμαστε μια υγιή τροφή. Αναφερθήκαμε πάρα πολύ και στο θέμα των ε, αντιβιωτικών. Το 1964 όταν αρχίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, στα 10.000 λίτρα γάλακτος που παραγόνταν τα 124 ήταν γεμάτα αντιβιωτικά. Τώρα έχουμε 2 λίτρα στις 10.000 και αυτό σημαίνει ότι με την πρόληψη τα τρόφιμα τελικά που φτάνουν στο τραπέζι μας ε, είναι ποιοτικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η πρόεδρος. Πώς να συνεχίσουμε. να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας από την Κανταβρία στην Ισπανία. Ελπίζω ότι κάτι θα μάθετε από τη σημερινή ακρόαση και θα πάρετε και μία ιδέα από τη σημασία του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον τομέα της ε, γεωργίας. Σας καλωσορίζουμε όλοι. Ο λόγος τώρα στον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ε, λίγες εβδομάδες ε, συνάντησα πολλούς εκπροσώπους από τους κοινοτρόφους ε, στην δική μου περιοχή, στην Καντάβρια και μου εξέφρασαν πολύ μεγάλες ανησυχίες γιατί βλέπουν νέες εμφάνισεις ευρουκέλωσης και φυματίωσης και έπρεπε να αυξηθούν τα κονδύλια για να για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Πριν λίγους μήνες απέφθηνα μία ερώτηση στην Κομισιόν για το θέμα αυτό και θεωρώ ότι στην απάντησή της ε, βρίσκεται το κλειδί όλων. Δηλαδή ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Και υπήρχε ε, τελικά ένα νέο συναγερμός για την εμφάνιση αυτών των όσων και θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Αλμάντσα να διπλασιάσει τις προσπαθίες του και πραγματικά να καθησυχάσουν τους κτηνοτρόφους που ε, υφίστανται πολύ μεγάλες ζημίες ότι θα αποζημιωθούν δεόντως. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα σε αυτή την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα διασφαλίσει ότι όλες οι ε, νόσοι θα αντικατοπτρίζονται στη βασική πράξη. Σας ευχαριστώ. Στην ε, πρόταση που έχουμε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ακριβώς αυτό, να καθορίσουμε ποιες αρρώστιες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και ποια ζώα. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ε, πράξεων κατεξοδότηση, αλλά νομίζω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει, οι κατάλογοι των ασθενειών θα πρέπει να υπάρχουν στην βασική νομική πράξη. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Τότε θα προσπαθήσω να συνοψίσω την ακρόαση που είχαμε σήμερα το απόγευμα. Ακούσαμε πολλά διαφορετικά θέματα. Καταρχάς, το θέμα του εθνικού καθεστώτος, πώς θα πρέπει να λύσουμε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ε, μεταξύ των διαφόρων περιφερειών στην Ευρώπη. Ε, θέλουμε κοινή ενιαία αγορά, θέλουμε ε, όμοιες προϋποθέσεις, αλλά ξέρουμε επίσης ότι οι φυσικές, ε, κλιματικές ε, συνθήκες αλλά και οι παραδόσεις, ε, οι πολιτιστικές προϋποθέσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τα εθνικά σχέδια και το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Και έτσι επανερχόμαστε στο θέμα της Πολωνίας. Η Πολωνία έχει μια παράδοση. Εγώ ίδια πριν 25 χρόνια είχα, είχα κάνει ρεπορτάζ για την πολωνική αγορά. Και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης έχει ένα είδος ε, αγορών ε, ε, ζωντανών ζώων. Στη Σκανδιναβία δεν υπάρχει η παράδοση αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει στη Ρουμανία ή την Ισπανία. Αλλά το θέμα είναι, είναι αυτό εθνικό ζήτημα ή είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. άσχετα από το πόσο νόμιμες ε, είναι αυτές οι αγορές. Επανερχόμαστε λοιπόν ε, στη συζήτηση. σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην καλή διαβίωση των ζώων και την ομοθεσία που μας λείπει και που δεν συμπεριλαμβάνονται ακριβώς στο συγκεκριμένο κανονισμό. ειλικρινά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες ε, στον ε, παρόντα κανονισμό, διότι θα παραγίνει πολύπλοκος. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την εφαρμογή και να έχουμε έναν κοινό βασικό νόμο για την προστασία των ζώων στο σύνολο της Ευρώπης, ώστε οι συνθήκες να είναι ίσες για όλους, αλλά ώστε και οι αγρότες στις διάφορες περιφέρειες ε, να έχουν λογικές συνθήκες ανταγωνισμού. Ε, σήμερα υπάρχουν κάποιοι ε, γεωργοί οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες ενώ σε άλλα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν νόμοι για την ε, προστασία των ζώων, για την καλή διαβίωση των ζώων και αυτό δημιουργεί μια καταστροφική κατάσταση. Και αυτό συνδέεται και με το όλο πρόβλημα της ανθεκτικότητας ε, στα αντιβιωτικά στο πακέτο που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, θεωρούνται και κεντροευρωπαϊκή απειλή για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, αλλά στην πραγματικότητα η κατανάλωση και κατάχρηση των αντιβιωτικών συνδέεται με τις εντιμικές ασθένειες. Αυτές που δεν έχουν ε, καταγραφεί ως μεταδοτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι ασθένειες ε, οδηγούν τους αγρότες σε οικονομικά και πρακτικά προβλήματα ε, καθώς και την κατάχρηση των αντιβιωτικών. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τη σχέση ανάμεσα σε όλες αυτές τις αντίθετες τάσεις ε, και να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Να ρωτήσω άλλη μία φορά, υπάρχει καμιά αντίρρηση στη σύνοψη που έκανα. Όχι. Όλοι σιωπούν. Ελπίζω. Ε, πρόεδρε, ρωτήσατε αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Θα πρέπει να συμφωνήσω όσον αφορά τα διάφορα πρότυπα και τι ε, προσεγγίσεις απέναντι στην καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Γκέκλε είναι ακόμα εδώ. Ε, μίλησε για το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κουνάβια, του ασβού. Ε, Έχουμε και την φυματίωση των βοηδών και υπάρχουν άλλα μέρη όπου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπου δεν αποτελεί προτεραιότητα η καλή διαβίωση των ζώων και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συζήτηση. Όμως, Ομολογώ ότι όταν άκουσα τα της των ζώων στις παράνομες αγορές κλπ. Το σημαίνει στην Πολωνία, στην Αγγλία, στην Βόρειο Ιρλανδία. Μου σκόρχε τρίχα. Και δεν είναι μόνο θέμα προστασίας των ζώων. Εγώ πιστεύω ότι τα ζώα πρέπει να διακινούνται ως σφάγια και όχι ζωντανά. Νομίζω συμφωνούμε όλοι με αυτό. Για να φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να θεσπίσουμε μία αρχή, η οποία θα ισχύει παντού σε όλες τις χώρες. Πρέπει επίσης αυτή η ελάχιστη νομοθεσία να εφαρμόζεται και να επιτηρείται σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούν οι Βρυξέλλες να ασχολούνται με την εφαρμογή της νομοθεσίας στην κάθε χώρα. Δείτε τι έγινε στο παρελθόν με την προστασία των ζώων, με τις απαραίτητες συνθήκες του στάβλου, τα πτυνοτροφία. Μετά δόθηκαν ένα σωρό εξαίρεσεις, παρεκκλήσεις. Κάποιοι δεν εφαρμόζουν τίποτα. Οπότε Εν τέλει διερωτώ Τα κράτη-μέλη, τα σωστά κράτη-μέλη που έχουν και τα υψηλότερα κόστη, μέχρι πότε θα δέχονται προϊόντα από τις γειτονικές χώρες που κάνουν ό,τι καπνίσει. Είναι ένα από τα πολλά ερωτήματα. Ε, δεν είμαι κατά της βελτίωσης της νομοθεσίας, αλλά ξέρετε εγώ έρχομαι από αγροτική περιοχή και θέλω διασφαλίζουμε ότι τα ζώα τρώνε και πίνουν πριν καν από εμάς. Έτσι κάνουμε στην περιοχή μου. Οι περισσότεροι αγρότες, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι αυτό κάνουν σε όλη την Ευρώπη. Τώρα υπάρχουν διάφορες ιστορίες και εδώ και εκεί και μπορεί να έχουν γίνει και στη δική μου περιφέρεια. Δεν το αποκλείω καθόλου. Κάποιοι να κακομεταχειρίζονται τα ζώα για κάποιο λόγο. Για αυτοί πρέπει να πεταχθούν. Λοιπόν, να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η συγγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλό συγκερασμένη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, είτε μιλάμε εντός μιας χώρας, είτε μιλάμε για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η ελεύθερη αγορά για τα ζωντανά ζώα, τα ζωικά προϊόντα κλπ. εξαρτάται από τον καλό έλεγχο των πιο επικίνδυνων ασθενειών. Και όσον αφορά τα τρόφιμα, να έχουμε τέτοιο έλεγχο της ζωής του ζώου, ώστε τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά να μην μπορούν να μεταφερθούν, για παράδειγμα, στους καταναλωτές. Συναντούμε πολλά ανθεκτικά βακτήρια στο κρέας των πουλερικών στην Ευρώπη και φαίνεται ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό σκάνδαλο. Υπάρχει άλλη μια ε, άλλη μια ερώτηση που θέλω να κάνω, θέλω να επαναλάβω. Στην πρότασή μου άγρια ζώα είναι όλα τα ζώα που δεν έχουν ιδιοκτήτη. για τα οποία δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος άνθρωπος. Και έτσι καλύπτεται και ε, ο σκύλος, ο αδέσποτος στο δρόμο και ε, η λύκη στα δάση. Δεν υπάρχει σαφής νομικός ιδιοκτήτης υπεύθυνο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο ορισμός που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε να σας ευχαριστήσω όλους ε, θερμά, όλους τους ομιλητές που ήρθαν ε, στις Βρυξέλλες ε, και που μας έδωσαν τόσες πληροφορίες και σας υπόσχομαι ότι θα κρατήσω τις φωτογραφίες από την Πολωνία, αλλά θα χαιρόμουν πολύ αν δεν χρειαζόταν να τις κοιτάω και ελπίζω να μην δούμε και άλλες τέτοιες. Ελπίζω δηλαδή να προοδεύσουμε στο θέμα αυτό. Με μια νομοθεσία που να επιτρέπει στα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αξιοπρεπή ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 9 με ψηφοφορίες μεταξύ άλλων πάνω στον προϋπολογισμό και τον κανονισμό που συζητήσαμε σήμερα. Όπως είπε κάποιος, ο προϋπολογισμός είναι σημαντικός, αποτελεί όμως μια μικρή τραγωδία στη σύγχρονη Ευρώπη, τη στιγμή που θέλουμε να πετύχουμε τόσα πολλά με τόσο λίγα χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.